Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε που με βοηθάτε. Η πρόεδρός μας απουσιάζει. Έχω λοιπόν την ευχαρίστηση και την τιμή να προεδρεύσω εγώ. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση και υπομονή. Θα ξεκινήσουμε με τις ε, ψηφοφορίες και εν συνεχεία θα έχουμε δύο ακροάσεις. Έχετε καταρχάς την έκθεση από τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές χθες το απόγευμα. Έχουμε λοιπόν τα πρακτικά από τις ε, δύο προηγούμενες συνεδριάσεις των συντονιστών της 9ης Νοεμβρίου και της 22ης Νοεμβρίου. Σας δόθηκαν λοιπόν τα πρακτικά που συνοψίζουν ε, τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων των συντονιστών και θεωρούν ότι αυτά εγκρίνονται αν δεν λάβουμε κάποια αντίρρηση μέχρι το τέλος συνεδρίασης. Σας προτείνω να περάσουμε ευθύ αμέσω στις ψηφοφορίες. Ας κάνουμε πρώτα μία δοκιμή για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα και αν είμαστε όλοι εδώ παρόντες. Να επιβεβαιώσουμε επίσης ότι δεν υπάρχει υπεράριθμος από καμία πολιτική ομάδα. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ πολύ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ψηφίσατε όλοι. Λείπουνε δύο, λείπει ένας ακόμα. Ένας από ό,τι φαίνεται δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Ποιος δεν ψήφισε. Εγώ ψήφισα. Πολύ ωραία, μάλιστα. Πολύ ωραία, δεν υπάρχει υπεράριθμος από καμία πολιτική ομάδα λοιπόν. Πολύ όμορφα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ε, ψηφοφορίες και καταρχάς με την έκθεση της κυρίας Ντεμόντε όσον αφορά την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Περιμένουμε να καθίσει και ο Βήμα. Έκθεση Ντεμόντε λοιπόν, συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 18, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική. Συμβαστική. του εντάξει, ρωτάει ο πρόεδρος. Πολύ ωραία. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 τώρα, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, πολύ ωραία, κάνα πρόβλημα. Άρχεται η ψηφοφορία για τροπολογία 42. Υπάρχει ένας ο οποίος αργεί να ψηφίσει από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραία πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44 τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 46 καταπίπτει και περνάμε στη 47 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 58, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Και όντω εγκρίνεται. Μία ψήφο διαφορά, 20 υπέρ, 19 κατά. Περνάμε σωμαστική 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 56 άρχιτη ψηφοφορία. πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τροπολογία 3. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψοφορία ηλεκτρονικά. Άρχιτη ψοφορία Πέρας. 33 υπέρ, 2 κατά και 5 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία και συγχαίρουμε την κυρία Ντεμόντε. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Έκθεση Μαρινέσκου για την προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Έκθεση λοιπόν του κυρίου Μαρινέσκου, όπως είπαμε. Ξεκινάμε τη ψηφοφορία. Συμβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 τώρα υπέρ. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική υπαριθμών 3 εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται η 14. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά, άρτη ψηφοφορία για τροπολογία 16. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική 5 εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Qui 34 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 34. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να, να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 22-19 εγκρίνεται. 44 υπέρ. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Περνούμε απευθείας... Στην συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέσει. Εγκρίνεται. Επομένως, ή 52, 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ζητείτε ηλεκτρονική ψήφος και έρχεται. Πέρας. και απο... απορρίπτεται. Λάθος έκανα εγώ, απορρίπτεται. Μάλιστα. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται πράγματι. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση παρακαλώ για την 55 άρχεται η ψηφοφορία. Για την 55 λέμε έτσι, λέει ο πρόεδρος. Πέρασε. Απορρίπτεται. 56 τώρα. Υπέρ. Κατά. Και εδώ να επαληθεύσουμε. Για την 56 παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επομένως 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 60 να ηλεκτρονική ψήφος στην 60 λοιπόν άρχεται πέρας Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική 12 εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, άρα είμαστε στη συμβαστική δεκατρία υπέρ. Αποχές λέει ο πρόεδρος από το υπέρ. Μετά το κατά. Εγκρίθηκε μπαστιτός 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 93. Συμβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές ή 103 απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχής. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κρίνεται. Συμβαστική 16 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία στην 120. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 με συγχωρείτε υπέρ, κατά, εποχές, να επαληθεύσουμε την 128 παρακαλώ. Πέρας, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, Νομίζω ότι έχουμε την ίδια πλειοψηφία, αλλά να επαληθεύσουμε την 129. Πέρας. Και ακριβώς η ίδια, 21-20 τώρα. το εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και επομένως περνούμε στην 145 υπέρ κατά αποχές η 145 εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά απορρίπτεται η 149, 150 υπέρ κατά αποχής να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας εγκρίνεται. 151 είναι υπέρ κατά εποχή εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μου ζητούν επαλήθευση ε, την 152 παρακαλώ πέρασε Εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τελική ψηφοφορία. Άρχεται παρακαλώ η ψηφοφορία. Και πέρας. 38 έναντι τριών και μηδέν αποχές συγχαρητήρια στον κύριο Μανέσκου. Πάμε στην τελευταία μας ψηφοφορία. Μια σύσταση για τις ε, αερομεταφορές με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγητής η κυρία Γκρίφιν. Με ηλεκτρονική ψήφο λοιπόν Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Θαυμάσια. 38-0 με τρεις εποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκρίφιθ. Επομένως ολοκληρώσαμε τις ψήφους. Και περνάμε τώρα στο hearing, λέει ο Πρόεδρος. Cette audition Σχετικά με τα τέλη της κυκλοφορίας ε, στο δίκτυο το οδικό μαζί με τα ηλεκτρονικά διόδια και τα υπόλοιπα. Bien, alors. Λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, συνάδελφοι, τώρα που ησυχάσαμε λίγο μετά την ψηφοφορία, να περάσουμε στην ακρόαση για το πάνελ όπως και για τα μέλη θα λειτουργήσουμε όπως και χθε. Δεν ξέρω αν έχω την ίδια εξουσία όπως και άλλοι πρόεδροι. Σας παρακαλώ όλοι να μείνουν αυστηρά εντός των ορίων που θα έχουν για τις τοποθετήσεις τους. Τώρα η ακρόαση μετά την χθεσινή ε, ασχολείται με τα οδικά τέλη το οποίο είναι σημαντικό θέμα διότι προσπαθούμε να κατανείμουμε το άχθος του οδικού δικτύου να καταπολεμήσουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν να εφαρμόσουμε την ε, αρχή του ότι ο χρήστης αναλογικά θα πρέπει να αναλαμβάνει το άκθος και ένα πλαίσιο τεχνικών ζητημάτων, εν πάση όλα αυτά που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση των υποδομών του οδικού δικτύου και του τρόπου με τον οποίο αυτό το σύστημα παράγει έσοδα. ή δαπάνηση. Εν πάση περιπτώσει το οδικό δίκτυο είναι ο βασικότερος άξονας μεταφοράς εμπορευμάτων και ανθρώπων αυτή τη στιγμή, είτε μας αρέσει είτε όχι. Να παρουσιάσω και τα μέλη του πάνελ που έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας, τον κύριο Γκαμπριέλε Μπενεντέτο, που είναι διευθύνων σύμβουλος της Τελεπάς του ηλεκτρονικού στήματος διοδίων στην Ιταλία, τον κύριο William Τόντζ, διευθύνοντα σύμβουλο της Transport and Environment, την κυρία Λοριάν Κρίντ από την Ομοσπονδία του Αυτοκινήτου, τον κύριο Λεμπεντά, International Road Union, τον κύριο Λόχμαν όπως και τον κύριο Διονέλη που εκπροσωπεί την ΕΣΕΚΑΠ European Association of Operators of Toll Road Infrastructures. Θα τις ακούσουμε με τη σειρά. Θα δώσω και το λόγο στους διάφορους ε, υπόλοιπους φορείς. Ε, θυμίζω σε όλα τα μέλη ότι έχουν 7 λεπτά. Υπάρχει χρονόμετρο το οποίο θα τους παρακολουθεί. Παρακαλώ και πάλι να είστε εντός των περιθωρίων του χρόνου που σας δίνουμε για να έχουμε το μέγιστο χρόνο για τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μπενεντέτο από το σύστημα ηλεκτρονικών διοδίων της Ιταλίας. Παρακαλώ κύριε Μπενεντέκτο. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω κάποιες διαφάνειες για να σας παρουσιάσω το Telepass που όπως είπατε Πρόεδρε είναι το σύστημα πληρωμής οδικών τελών, διοδίων δηλαδή, Είμαστε ηγέτη στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Έχουμε 6 εκατομμύρια πελάτες μέσω 11 εκατομμυρίων τίτλων πληρωμής. Δηλαδή έχουμε περί το 30% της αγοράς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα διόδια. Αναέτος κάτι λιγότερο από 6 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλος εργασιών και εκπροσωπούμε ένα, μια μεγάλη αλυσίδα φορέων που σχετίζονται με την ε, υποδομή του οδικού δικτύου και ως τέλεπας έχουμε μια ηγετική θέση γιατί ξεκινώντας από την Ιταλία έχουμε καλύψει και άλλα σημεία της Ευρώπης ε, προσπαθώντας να καλύψουμε το δύσκολο πρόβλημα της διαλειτουργικότητας ε, που σήμερα βλέπουμε πλέον να οθείται να υπογραμμίζεται στην οδηγία. Εμείς ε, ελπίζουμε να πλουστευτούν τα πράγματα γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα διάφορα οχήματα ε, με εννέα μηχανήματα να κυκλοφορούν προκειμένου να επικοινωνούν μεταξύ των συστημάτων. Υπάρχει λοιπόν με σημαντική προστιθέμενη αξία που μπορούμε να επιτύχουμε μέσω της διαλειτουργικότητας. Οπωσδήποτε υπάρχει ένα θέμα κόστους για τον τελικό χρήστη αλλά υπάρχει και ένα θέμα ε, για τους φορείς που πρέπει να αναπτύξουν πολλά και διαφορετικά πρότυπα επί τη αγορά. Για το λόγο αυτό, η τροποποίηση των, ε, της προθεσμίας των 24 μενών της προηγούμενης εκδοχής οδηγίας ε, είναι θετικό, διότι είναι ελκυστικό για τους φορείς και δεν χάνουμε και το καθεστώς του ή ETS provider, αν ακούσαμε καλά. Ήταν ε, σημαντικό που είχαμε on-board unit, δηλαδή δορυφορική σύνδεση μηχάνημα που βρίσκεται μέσα στο όχημα, που έχει πολύ μεγαλύτερη, πολύ ευκρινέστερη εμβέλεια και, είναι, και αντιπροσωπεύει το 80% της αγοράς αυτή τη στιγμή για να διαβάζει ακριβώς τα ηλεκτρονικά διόδια. Πρόκειται για το πρότυπο αυτή τη στιγμή της αγοράς. Εκτιμούμε τα όσα έλαβαν χώρα στην, στα πλαίσια της αναθεώρησης οδηγίας προκειμένου να επιτηρηθούν τα τεχνολογικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους φορείς ε, των ε, κρατών μελών. Θα επανέλθω σε αυτό αλλά ήθελα μια στιγμή να υπογραμμίσω τις πτυχές εκείνες στις οποίε κατά την άποψή μας χρειάζεται ακόμα λίγη δουλειά. Πρέπει να μην υπάρχουν εμπόδια εισόδου όταν ε, ένας φορέας όπως εμείς προσπαθεί να πάει σε άλλες διεθνείς αγορές. Υπάρχουν επίσης κάποιες ε, δυσκολίες όπου έχουμε τελείως διαφορετικά έντυπα ή έγγραφα που μας ζητούνται από τους φορείς του συστήματος διοδίων. Διαφορετικές διαδικασίες πιστοποίησης της τεχνολογίας, ε, της τεχνολογίας, τα πρότυπα, γλωσσικά, πάρα πολύ συχνά τα αγγλικά δεν είναι καθόλου η πρώτη γλώσσα των όσων μας ε, παραδίδουν αυτά τα έντυπα, και πολύ διαφορετικά συστήματα τελών, αποζημίωσης και αμοιβή στα διάφορα κράτη. Κάθε πάροχος ε, θα πρέπει να έρθει σε διεπαφή με όλα αυτά τα διαφορετικά συστήματα σε διαφορετικές γλώσσες και με διαφορετικά πρότυπα. Και επομένως το τεχνολογικό ζήτημα θα έχετε καταλάβει ήδη από την παρουσίασή μας, μου, είναι θέμα κλειδί. και δεν δίδεται μέσω των παρατημάτων παρκές ειδικό βάρος ακριβώς στο τεχνολογικό επίπεδο. Εμείς το 99,7% των εσόδων μας το διαχειριζόμαστε με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως χρεώσεις δηλαδή των δύο που γίνονται στο δικό δίκτυο πρέπει να αποφύγουμε συγκρούσεις ή δυσλειτουργίες με τα υφιστάμενα συστήματα. Ο κόσμος πηγαίνει προς την δορυφορική τεχνολογία, όλοι την αγκαλιάζουμε ενθουσιοδός, με ηγέτιδα φυσικά τη Γερμανία. Οποιαδήποτε μεταβατική φάση ε, απειλεί την επιτυχία του παρόντος συστήματος του 5,8 μεγακύκλων, γίγακύκλων με θεωρείτε. Έχουμε και το θέμα των διασυνοριακών ανταλλαγών ε, δεδομένων που μας επιτρέπουν να έχουμε και μία επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιώντας ακριβώς τη λειτουργικότητα μέσω της τεχνολογίας. Ε, είναι σαφής ότι σε κάθε χώρο ο ρόλος του φορέα του συστήματος, ε, του φορέα ίσπραξη των διοδίων κτλ. είναι τελείως διαφορετική. Η ιεράρχηση μεταξύ τους και η διάρθρωση μεταξύ τους. Θα χρειαστεί λοιπόν και μία... ο καθορισμός κάποιων προτύπων Διότι τα, οι χώρες που χρησιμοποιούν καθαρά εγχώριο σύστημα είναι αδιανόητο ότι να σκέφτονται ότι θα μπορούσαν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις της διαλογικότητας ε, και να μείνουν απομονωμένες. Ε, ε, η θέση λοιπόν ομοιόμορφων προτύπων σε όλο το εύρος του συστήματος είναι ένα από τα σε μια κλειδιά για μας. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. <coughs> Σας ευχαριστούμε κύριε Μπενεντέτο. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κρίντα, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Κυρία Κρίντα, έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εμεί στην FAI Region 1 προσωπούμε 37 εκατομμύρια μέλη στον τομέα της κινητικότητας. Αυτό λοιπόν συνάντη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος ε, στο περιβάλλον για να διευκολύνουμε τις μεταφορές και τους χρήστες στα ταξίδια του. Μας ανησυχούν οι προτάσεις που ε, προσπαθούν να εφαρμόσουν ε, μονομερείς, αν θέλετε, λύσεις σε ήδη υφιστάμενα εθνικά σχέδια και μας ανησυχούν ότι τα στοιχεία που εντοπίζονται και τα προβλήματα που έχουμε δεν ε, επιλύονται. Ο πρόεδρο ε, τονίζει στην κυρία ότι θα πρέπει να μιλάει λίγο πιο αργά, εάν θέλει να την παρακολουθούν οι δερμηνοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ήδη μεγάλη το φορτίο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν θα επιληθούν από την πρώτη σε και ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι το καλύτερο για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα. Και το πρώτο λοιπόν σημείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να γίνεται πληρωμή ανά Βλέπετε ότι 82% των φόρων και των επιβαρύνσεων ήδη έχουν να κάνουν με τη χρήση του δρόμου. Όσο πιο πολύ οδηγεί κανείς, όσο πιο πολύ πληρώνει κανείς τέλη ε, φόρους και αυτό είναι ήδη έτσι σήμερα. Η πρόταση λοιπόν να αλλάξουν τα συστήματα για να υπάρξει χρέωση ανά χιλιόμετρο είναι μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το μελέτη που της Επιτροπής υπολογίζει περίπου 1,2 δις επιπλέον κόστος για το σύστημα το οποίο θα το καλύψουν τελικά οι χρήστες. Άρα το συμπεράσμά μας είναι ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα χρήσης, ανα, μάλλον πληρώμες αναχρήσεις. πιστεύουμε ότι τα εθνικά συστήματα είναι καλύτερα και το κόστος, ε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα το ε, πάρουν πάνω τους οι οδηγοί, οι πολίτες. Και αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντικτύπωση σε όλη την κοινωνία. Ούτε αναλογικότητα ούτε επικορικότητα τηρούνται. Δεύτερο στοιχείο σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση για τις υποδομές. Οι μελέτες μας καταδεικνύουν ότι το 2013 είχαμε 286 ε, δισεκατομμύρια έσοδα στην Ευρώπη των 27 σε ό,τι αφορά τα κτίρια και σε ό,τι αφορά τη συντηρήση των δρόμων. Μιλάμε για 108 επιπλέον της ε, ε πλεόνασμα σε τα έσοδα. Έχουμε 203 εκατομμύρια που πληρώνουμε από τα αυτοκίνητα και 93 για τις υποδομές. Και αυτό καταδεικνύει, βλέπετε στο γράφημα στο κάτω μέρος της διαφάνειας, ότι οι επενδύσεις στην υποδομές έχουν μειωθεί από 1,1 του ΑΕΠ το 99 σε λιγότερο από 1,8 του 2010. Άρα, υπάρχει ένας μηχανισμός ανακατανομής όπου οι οδηγοί συμβάλλουν στον εθνικό υπεροπολογισμό. Η ευρωπαϊκή πρόταση ε, προβλέπει καταμέτρηση και ε, των ε, επενδύσεων και σημαίνει υποχρεώσεις, αλλά υποχρεώσεις αυτές δεν εγγυώνται ίσως τη συντήρηση. Το συμπέρασμα μας λοιπόν είναι ότι Ήδη η ποικιλία των εθνικών μέτρων και επιβαρύνσεων φροντίζει για την συντήρηση και τις υποδομές και συμφωνούμε ότι αν δεν τηρούνται καλά οι υποδομές αυτό επηρεάζει και το περιβάλλον και την ασφάλεια και είναι αποδεδειγμένο ότι η επιδιόρθωση είναι πιο ακριβή από τη συντήρηση των δρόμων. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά για την βελτίωση των υποδομών. Ένα άλλος στόχος είναι να δώσουμε όθηση στα καθαρά οχήματα. Και εδώ ε, γίνεται διάκριση στις τιμές σε ό,τι αφορά το επίπεδο των εκπομπών των οχημάτων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας υπενθυμίσουμε ότι η φορολόγηση στα κρατημέλη ήδη ε, βασίζεται στις εκπομπές και προωθούνται τα πιο καθαρά οχήματα από τις κυβέρνησεις. Αυτό αλλάζει φυσικά ως τεχνολογική ε, ω τεχνολογικό ε, κλάδο. Παλιά ήταν ντίζελ, τώρα τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα παραλλάζουν και τα επιστημονικά στοιχεία. Και ήδη τα καθαρά οχήματα προωθούνται από πολλέ νομοθεσίε ε, για τις πραγματικές εκπομπές για να εξασφαλίσουμε ότι πραγματικά πετυχαίνουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Δεν είμαστε από όλοι βέβαιοι τι θα σημαίνει αυτή η νέα αυτό το νέο επίπεδο και είναι και ένα ελαστικό αυτό το μέσο και ουσιαστικά διακυβεύει τις μεταφορές στην Ευρώπη για την πρόταση τώρα σε ό,τι αφορά τους παράγοντες ε, συμβατότητας για την καταμέτρηση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό δεν επιτρέπεται από το υφιστάμενο πλαίσιο και θέλουμε... Η πρόταση θέλει πιο μεγάλη υποστήριξη των καθαρών οχημάτων. Ω εκπρόσωπο των χρηστών, όμω, θα πρέπει να σα πω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, εναλλακτικές, βιώσιμε συναλλακτικέ. Ε, για τους ε, χρήστες, ε, για παράδειγμα, στις, ε, στην Ήπεθρο. Και υπάρχει και ο κίνδυνος να στραφεί η κυκλοφορία τελικά στις μεθόδρες αρατηρίας. Τι πιστεύουμε λοιπόν, πού πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί η πρόταση μετά από αυτά που σας παρουσιάσαμε. Ναι, υπάρχει ποικιλία στα εθνικά συστήματα, στην φορολογία και μπορεί να είναι δύσκολο να περάσει κανείς τα σύνορα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποια μέτρα ενδεχομένως να έχουν διακριτική επίπτωση σε κάποιες εθνικότητες και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προβλέπει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση βάσει εθνικότητας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή προστατευμένη αξία θα πρέπει να διατηρήσει την διαλειτουργικότητα των ε, συστημάτων σε ό,τι αυτή την χρήση ανά την πληρωμή αναχρήση. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα συστήματα θα σέβονται πλήρως ε, τη νομοθεσία για προστασία των δεδομένων και οποιαδήποτε στοιχεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς ε, πέραν από αυτούς για τους οποίους προορίζονται κλείνοντας ε. η πρόταση Όσο έχει θεωρώ ότι θα έχει θεωρώ ότι ούτε θα πετύχει όσα υποτίθεται θα πρέπει να πετύχει για υποδομέ και για τι μεταφορέ και θα επιβαρύνει πιο πολύ του χρήστε. Και βλέπουμε ότι ήδη οι οδηγοί επιβαρύνονται υπερβολικά για τη διατήρηση των υποδομών και πιστεύουμε ότι δεν θα τηρηθούν και οι αρχέ τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα βάσει του άρθρου 91 τη συνθήκη. Θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ βιώσιμε για τον κόσμο. Καλούμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να καταρτήσει μια ισορροπημένη τέτοια έκθεση σε ό,τι αφορά την κινητικότητα που αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει το, ο κ. Στότς, ε, ε για τα θέματα περιβάλλοντος και μεταφορών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η T&E Transport and Environment είναι μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις που ασχολείται με τις οικολογικές καθαρές μεταφορές. Το ζήτημα της οδικής τιμολόγησης μας έχει απασχολήσει ήδη από τη δεκαετία του 90 και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε την παρουσίαση αυτή για τα οδικά τέλη, βλέποντας λίγο πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Από το 1999, όπου είχαμε την πρώτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ένα ολόκληρο κατάλογο κρατών, με τελευταίο το Βέλγιο και έπειτα τις κάτω χώρες που έχουν εισάγει ηλεκτρονικά συστήματα τελών χρήσης ε, οδικών δικτύου. Αυτό το οποίο έχουμε μάθει λοιπόν τελευταία χρόνια είναι ότι αυτή η οδική τιμολόγηση έχει κάποια πλεονεκτήματα. Αυτό έχει να κάνει με το ότι προωθούνται περισσότερο τα καθαρά οχήματα, καθότι υπάρχουν πιο ευνοϊκά μέτρα, πιο ευνοϊκά τέλη για τα οικολογικά οχήματα, δημιουργείται ένα πιο ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών και επίσης τα τέλη αυτά μπορούν να αποτελούν πολύ αποτελεσματικά μέσα προκειμένου να αυξάνονται οι πόροι του κράτους και να χρηματοδοτούνται οι οδικές υποδομές. Αν δούμε το σύστημα που έχει η Γερμανία, που είναι ένα από τα πιο πλήρη συστήματα στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι μολονότι μπορούν να υπάρχουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, από την άλλη ο αντίκτυπος δεν θεωρείται από οικονομικής πλευράς αρνητικός. Και νομίζω ότι Ορισμένοι συνάδελφοι ενδεχομένω να πούνε σήμερα ότι η οδική τιμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή. Κάτι δεν, αυτό δεν ισχύει στην πράξη όμω. Αν δούμε τώρα την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή είναι καλή. Από, από την άλλη υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωση. Τέσσερι συστάσει έχουμε να κάνουμε, οι οποίε έχουν να κάνουν με, με τι διαφορετικέ κατηγορίε οχημάτων. Να ξεκινήσουμε με τα βαρέα οχήματα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Έχει προκύψει τώρα μια κατάσταση όπου Πολλές χώρες ε, έχουν οδική τιμολόγηση για τα οχήματα αυτά, αλλά όσον αφορά την κάλυψη του κόστους ε, που προκαλούν τελικά τα φορτηγά, καταστροφή του δικού δικτύου, η ατμοσφαιρική ρήπανση, πάλι η κάλυψη αυτού του κόστους προκαλούν δεν είναι πλήρης. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του κόστου το οποίο μετακυλείται στου ε, υπόλοιπου πολίτε, στην κοινωνία. Σε εσά και σε μένα δηλαδή. Είμαστε πεπισμένοι λοιπόν εμεί ότι θα ήταν πολύ καλύτερο και για τους χρήστες αλλά και για τους ρηπαίνοντες να προχωρήσουμε σε ένα άλλο σύστημα το οποίο θα προβλέπει πρώτον ότι θα πρέπει να μπορούμε να εφαρμόσουμε ουσιαστικά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σταδιακή πάυση χρήσης της Ευρωβινιέτας καθότι στην περίπτωση αυτή άλλοι καταβάλουν το κόστος το οποίο θα πρέπει να καταβάλουν τα φορτηγά το εξωτερικό κόστο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι μέρο του εξωτερικού κόστου θα πρέπει να πάει σε τμήμα τη οδική τιμολόγηση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ομοιόμορφο σύστημα παντού στην εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορούμε τελικά το εξωτερικό κόστο να το εισάγουμε εντελώ στο σύστημα οδική τιμολόγηση. Να καλύπτεται πλήρω δηλαδή από το σύστημα οδική τιμολόγηση. Α περάσουμε τώρα σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ξέρετε ότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε στο τομέα των μεταφορών. Και οι οδικές μεταφορές, ιδίω οι οδικές εμπορευματικέ μεταφορές, συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στι ε, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό το πρόβλημα είχε αυξηθεί από τι αρχέ του 1990. Τώρα, το πρόβλημα με τα φορτηγά είναι ότι δεν έχουμε ακόμα πολλά μέσα, πολλά φορολογικά μέσα, προκειμένου να δίνουμε κίνητρα στη χρήση οικολογικών φιλοπεριβαλλοντικών φορτηγών. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιήσουμε την οδική τιμολόγηση, τα τέλη δηλαδή χρήση του δικού δικτύου, προκειμένου να δώσουμε κίνητρα φορολογικά στι επιχειρήσει οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν οικολογικά φορτηγά. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να δώσει νέα σε αυτή την αγορά και στηρίζουμε από αυτού την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτων. όσον αφορά τα μικρότερα φορτηγά. Θα έχετε δει στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, αλλά και σε άλλες χώρες, ότι έχουμε φορτηγά μικρότερου μηγέθους, τα οποία, τον οποίο ο αριθμός έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο είναι εύχριστα τα οχήματα αυτά, αλλά επίσης έχουν μία σειρά από ρυθμιστικά πλεονεκτήματα, καθότι δεν υπάγονται σε πάρα πολλούς κανόνες που ισχύουν για τα μεγάλα φορτηγά. Δεν ισχύουν οι κανόνες ταχογράφου για αυτά και δεν ισχύουν πολλοί άλλοι ρυθμιστικοί περιορισμοί. Γι' αυτό το λόγο προωθούνται αυτή τη στιγμή από πάρα πολλέ μεταφορικές εταιρείε. Θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει να καλυφθούν και τα μικρά αυτά φορτηγά από το σύστημα οδικής ετοιμολόγησης. Είδαμε για παράδειγμα ότι η απουσία οδική τιμολόγηση για τα ελαφριά αυτά φορτηγά οδήγησε στο Βέλγιο σε μία αύξηση τη χρήση κατά 20% τελευταία χρόνια. Θεωρούμε λοιπόν ότι και αυτά θα πρέπει να υπαχθούν όπω και τα βαρέα φορτηγά στο σύστημα οδική τιμολόγηση. Όσον αφορά τώρα τα επιβατικά οχήματα, τρία πράγματα θέλω να σα πω. Πρώτον, οι βινιέτε δεν είναι αποτελεσματικές, εισάγουν η διακριτική μεταχείριση και όπω είπα πριν από λίγο, οπουδήποτε έχουν χρησιμοποιηθεί, ουσιαστικά έχουν αναγκάσει τους ξένους να πληρώσουν. Αυτό συμβαίνει στι περισσότερες περιπτώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι αποτελεσματικό μέσο. Επίση υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ευρώπη. Αυτό μα κοστίζει μια ολόκληρη περιουσία. Ένα μέσο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τελικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι η οδική τιμολόγηση ανά χιλιόμετρο. Υπάρχουν πάρα πολλέ έρευνε που το δείχνουν αυτό. Θα είναι κρίμα να μην χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την χιλιομετρική οδική τιμολόγηση. Πρέπει να την ενθαρρύνουμε, θεωρώ. Τρίτη παρατήρηση. Η κινητικότητα τροποποιείται, μεταβάλλεται. Τα επόμενα 10-15 χρόνια θέλουμε να περάσουμε σε ένα πιο αυτοματοποιημένο ηλεκτροκινούμενο σύστημα μετακίνησης. Καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση αυτή οι μεταφορέ θα είναι πολύ πιο φτηνές και είναι πολύ πιο φτηνό και σαφώ λιγότερο δαπανερό να χρησιμοποιεί κανεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και πόσο μάλλον ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρί οδηγό, αυτόνομο, αυτοοδηγούμενο. Οι εξελίξεις αυτές, μολονότι έχουν ε, πολλές θετικές πτυχές, ενδεχομένως να δημιουργήσουν και κάποια προβλήματα σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων πλέον που θα έχουμε στους δρόμους μας και σε σχέση με τη μείωση των εσόδων που θα έχουμε από την ε, μείωση της φυρολογίας ε, στα καύσιμα. Νομίζω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί και με την τελευταία αυτή πτυχή και να δούμε πώ το πλαίσιο τη οδική τιμολόγηση θα μπορούσαμε να καλύψουμε και τη νέα αυτόνομη αυτή ηλεκτρονική κινητικότητα που μα περιμένει για το μέλλον. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Τότσα. Το λόγο τώρα έχει ο κύριο Ρεμί Λεμπεντά, ο οποίο εκπροσωπεί τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών, IRU. Κύριε Λεμπεντά, έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ε, καλημερίζω όλους σα. Ε. Είμαστε ε, η οργάνωση για τις οδικές μεταφορές. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των χειριστών λεωφορείων, ταξί, φορτηγών, μέσω εθνικών συνομοσπονδιών. Δεν χρειάζεται να σας πενθυμίσω τι σημασία έχουν οι μεταφορές ε, στην Ευρώπη και στον απορικό σκέλος φοιτητέρος. Σε ό,τι αφορά την Ευρωβινιέτα, από ό,τι φαντάζεστε το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για μας, γιατί αγγίζει τα συμφέροντα όλων των ε, φορέων της αγοράς. Πού θέλουμε λοιπόν να καταλήξουμε αυτή την πρόταση. Το κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τη διαφάνεια του αποτελέσματος. Και εδώ και χρόνια ζητάμε μια έκθεση επισκόπησης ε, σε ό,τι αφορά το κόστος υποδεμών και πιστεύουμε ότι μόνο με την σαφήνεια αυτή εγκάρσια θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστές ε, Συζητήσει και να λάβουμε σωστές αποφάσεις και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημοσιεύσει τέτοια έκθεση του χρόνου. Στο τρέχον πλαίσιο, σε ό,τι αφορά την ανάλυση της έκθεσης της Επιτροπής, βασιζόμαστε σε δύο επίπεδα. Χρήση των εσόδων και φορολόγηση. Ζητούμε λοιπόν ουδετερότητα σε ό,τι αφορά τα έσοδα σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά προϊόντων, σε ό,τι αφορά τους αυτοκινητοδρόμους και τι μεγάλε αρτηρίες, σε ό,τι αφορά την ρήπανση και τον θόρυβο. Ξέρουμε ότι τα ευρωπαϊκά φορτηγά καλύπτουν πάνω από 100% του κόστου του ήδη. Και δεδομένου ότι το δυναμικό αλλαγής ε, του τρόπου διακίνηση των μεταφορών από τον δρόμο σε άλλα μέσα μεταφορών είναι πολύ περιορισμένε οι δυνατότητε. Ε, η χρήση λοιπόν φορτηγών θα είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να μειωθεί λοιπόν το κόστος επένδυσης για τους α, ε, μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τις επιβατικές μεταφορές, ε, η επιβάρυνση είναι σε 15 και πάνω κράτη-μέλη και είναι πολύ διαφορετική εδώ η αγορά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και εδώ το αποτέλεσμα μεγαλύτερη φορολόγηση θα ήταν λιγότερα συλλογικά οχήματα, λεωφορεία, βαν και πιο πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους. Το οποίο είναι αντίθετο με την πρόσφατη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να δοθεί κίνητρο για τα λεωφορεία που θα είχε και σημαντικέ συνέπειε και για την ασφάλεια στους δρόμου και για το περιβάλλον σε κάθε περίπτωση αυτή η τιμολόγηση των οδικών μεταφορών δεν θα έπαιζε το ρόλο που θα έπρεπε ως κίνητρο για πιο καθαρές και πιο αποτελεσματικές μεταφορές. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτή η τιμολόγηση οδικών μεταφορών να μην παίξει το ρόλο του ασαντικίνητρου. Θα πρέπει να δούμε πως ε, κάθε τέλος θα εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Αν τα χρήματα πάνε στον γενικό προπολογισμό του κράτους, πρόκειται για φορολόγηση. Εμείς, από όσο καταλαβαίνουμε από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Και αν ε, πρόκειται για φόρο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και ως φόρος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση των προσόδων αυτών. Δεν είμαστε υπέρ ε, να χρησιμοποιηθούν στα κτίρια και στη συντήρηση των ε, δρόμων και για τους χώρους στάθμευσης. Ε, εμείς θέλουμε να πάμε πέρα από αυτά που θεωρούμε ότι συναποτελούν αυτή την αρχή. Γιατί είναι τόσο χαμηλό το δυναμικό αλλαγής χρήσης μέσων. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Θέλουμε να μειωθούν οι εκπομπές στην πηγή τους και να επιτρέψουμε στις οδικές μεταφορές να καταστούν σε θέση να μειώσουν τις εκπομπές. Θέλουμε τεχνολογία ε, καθαρών οχημάτων, εκπαίδευση, υποδομή, ITS, για να συνοψίσουμε τις προτάσεις μας να απαλλαγούν τα λεωφορεία και τα πούλμαν από το πλαίσιο αυτό προτείνουμε. Γιατί είναι σαφώς μέρη της λύσης και όχι του προβλήματος. Θα ήταν πραγματικά αντιφατικό να επιβαρυνθεί αυτή η δραστηριότητα και να υπαχθεί να μην υπαχθεί στους ε, νόμους της αγοράς και να δημιουργηθούν επιπλέον επιβαρύνσεις με την Ευρωβινέτα. Τουλάχιστον ως ε, αιτητικά οχήματα να αντιμετωπίζουν αντιμετωπίζονται στη χειρότερη περίπτωση τα ελεφόρια. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να έχουν την ελευθερία να επιλέξουν την ε, χρήση βινιέτα ή διοδίων, κατά πόσο θέλουν να επιβάλλουν τέλη ή όχι, σε ό,τι αφορά τη μετάβαση από γύρω κλάς ε, σε πρότυπα διοξιδίου του άνθρακου. Αυτό το καθορίζουμε, αλλά θέλουμε να γίνει αυτό με ε, τρόπο που να μην σημαίνει αλλαγή στα έσοδα και το κόστος αυτό να επηρεάσει την Ιρβινιέτα. Ε, η συγκεκριμένη χρήση των πόρων, το earmarking, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, προκειμένου να ε, διοχετευτούν αυτά τα έσοδα τελικά πάλι στι οδικέ μεταφορέ, να καταστούν πιο αποτελεσματικέ. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιβάρυνση λόγω συμφόρηση, ήδη πληρώνουν. Το κόστος αυτό ήδη εσωτερικοποιείται μέσω απώλειας δυνατοτήτων και μέσω φορολόγησης και συχνά. Να σας δώσω το παράδειγμα αυτό για τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Η Επιτροπή προτείνει να επιβαρύνονται και να φορολογούνται 2,5 φορές, ανα, τα, φορές σε σχέση με τα ιδιωτικά οχήματα. Ενώ ξέρουμε ότι ένα λεωφορείο μπορεί να αντικαταστήσει 30-35 οχήματα στους δρόμους. Και επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι τα πούλμαν και τα λεωφορεία αποτελούν μέρος της λύσης και του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο για 7 ε, λεπτά στον κύριο Λόχμαν από το CER. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μας δίνεται να εκφράσουμε την άποψη των ε, σιδηροδρόμων. Σχετικά με την χρέωση που είναι απολύτως ε, ρυθμισμένη σήμερα νομικά. Και είμαστε υπο, υποκείμενοι και σε αυτό που σήμερα αποκαλείται μερικές φορές ε, τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης λόγω της αυξημένης ζήτησης. Θα σας ε, αναφέρω κάποια στοιχεία που ανέφεραν και οι προηγούμενοι ε, ομιλητέ ε, μερικώ και κάποιε τάσει. Καταρχά, αν μου επιτρέψει και το σύστημα, α είμαστε σαφεί. Η ίδια η Εβραϊκή Επιτροπή με τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές το 2011 μίλησε για υποχρεωτική εσωτερικοποίηση των εξωτερικών κόστος μέχρι το 2020. Αυτό θα πρέπει να διέπει ως αρχή όλους τους ρηπαίνοντες, διότι θα πρέπει να βαρύνει τους ρηπαίνοντες και όχι την κοινωνία το κόστος αυτό. Και θεωρούμε ότι πρέπει αυτή η αρχή να εφαρμόζεται και να υλοποιείται. Αλλά με έκπληξη βλέπουμε ότι η Κομισιόν δεν ε, παρακολουθεί την φιλοδοξία της με υλοποίηση το οποίο ως αρχή αναφέρεται και στη συνθήκη. Ας έχουμε λοιπόν μια ισότιμη και δίκαιη απόφαση και μεταχείριση της ε, κοινωνίας σχετικά με τα συστήματα μεταφορών. Αφενός αυτό, αφετέρου. Κάποια δεδομένα που προκύπτουν από έρευνες. Μπορείτε να βρείτε και μια συνοπτική παρουσίαση εδώ στην είσοδο, με περισσότερα ακόμα δεδομένα από αυτά που σας δείχνω. Κατά μέσον όρο, σύμφωνα με τη μελέτη της CE Delft, το δικό δίκτυο καλύπτει μόνο το 30% του εξωτερικού κόστους, των επιχειρήσεων δηλαδή στο σύνολο των δικτύων. 70 έως 90% αν μιλήσουμε για τους αυτοκινητοδρόμους, αλλά εν πάση περιπτώσει σε καμία περίπτωση 100%. Είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτεί κανείς. Και επειδή αναφερθήκαμε σε κάποιες εξαιρέσεις ε, ε, χερσαίων μεταφορών, οι σιδηρόδρομοι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση ανάληψης αυτού του άχθους. Ε, δεν διακρίνονται δηλαδή από τα οχήματα όπως αυτοκίνητα και φορτηγά. Υπάρχει και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι τιμές αναφορές. Ε, θα πρέπει να ξεπεράσουμε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε δηλαδή το εξωτερικό κόστος και, με το, και τον τρόπο με τον οποίο το ε, καθιστούμε υποχρεωτικό. Επίσης θα πρέπει να αποχωρήσουν σταδιακά τα τέλη που βασίζονται στα διόδια. Θα πρέπει δηλαδή να εισαχθεί ένα σύστημα το οποίο να βασίζεται στην απόσταση που έχει διανυθεί. Όλα αυτά τα συστήματα διοδίων και τελών θα πρέπει να οδηγήσουν σε ένα πιο καθαρό σύστημα μεταφορών και θα πρέπει να είναι δίκαια για την κοινωνία. όπως και όλες οι προσαυξήσεις που υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτήσουν τους ε, διαδρόμους TNT. Η συστάσεις μας πέραν των όσων έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιλώ αναφορικά προς τη Λευκή Βίβλο που αναφέρει την υποχρεωτική ανάληψη των εξωτερικών κόστος, κόστος όλου του εξωτερικού με συγχωρείτε κόστου. Θα πρέπει δηλαδή κατα, καταρχάς να καταστήσει σε, όλες τις, ε, βασικές, σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες το τέλος που θα βασίζεται στην απόσταση. Θα πρέπει να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογή των εξαιρέσεων για να υποστηριχθεί το εξωτερικό κόστος Επίσης θα πρέπει να υποστηριχθούν τρόποι ώστε να υπολογίζεται αυτό το εξωτερικό κόστος για να υποστηρίξουμε τις καθαρές μεταφορές και θα πρέπει να εξασφαλίσουν άμεση χρέωση, άμεση ανάληψη του κόστους αυτού μέσω της μείωσης των εσόδων των διοδίων. Γιατί ακόμα και τα ηλεκτρον, οι ηλεκτρονικοί σιδηρόδρομοι που είναι απόλυτος καθαροί, καθαρό σύστημα μεταφορών, αυτή τη στιγμή επιβαρύνονται. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί η αρχή των καθαρών συστημάτων ως εξαίρεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Euh. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λόχμαν. Έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις, βλέπω. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Καλίστρατος Διονέλης, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση των Φορέων Εκμετάλλευσης Οδικών Υποδομών Διοδίων. Κύριε Διονέλη, έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και να καλωσορίσω και τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ. Η ΑΣΕΚΑΠΑ εκπροσωπεί ουσιαστικά όλους τους δρόμους, γέφυρες, σύραγγες στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να προσφέρουμε ποιότητα, ταχύτητα, ασφάλεια και γι' αυτό το λόγο βέβαια λαμβάνουμε και κάποια τέλη με τη μορφή διοδίων που αποτελούν ένα μέσο χρηματοδότησης για μας. Εμείς εκπροσωπούμε τις Εθνικές Ενώσεις των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε λοιπόν μια πανευρωπαϊκή ομοσπονδία η οποία παρτίζεται από τις Εθνικές Ενώσεις Εκμετάλλευσης των Υποδομών Διοδίων. Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή σταδιακής απαλλαγής από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Συμφωνούμε όλοι επ' αυτού και όσον αφορά τις οδικές μεταφορές βλέπουμε ότι πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να γίνουμε κοινωνίες πιο οικολογικές και να μα χειροκροτούν και οι πράσινοι τελικά, να μας επιθυμούν. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε δύο βασικέ αρχέ. Η αρχή ο χρήστης πληρώνει και η αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει. Όπου έχουμε εδώ πέρα ουσιαστικά μια εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Αν ισχύουν οι δύο αυτές αρχές, θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται και στην πράξη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Πρώτον, και θεωρώ ότι αυτό είναι πρωταρχική προτεραιότητα στην οδηγία όσον αφορά την Ευρωβινιέτα, να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα της χιλιομετρικής τιμολόγησης. Πρόκειται βασικά για το βασικό μέσο προκειμένου να εφαρμοστούν οι δύο αυτές αρχές επί των οποίων όλοι συμφωνούμε. Η αρχή ο χρήσης πληρώνει και η αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει. Επίσης, μα δίδεται στην πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δυνατότητα να διατηρήσουν ορισμένα κράτη, ορισμένες περιφέρειες, την τιμολόγηση βάσει της χρονικής διάρκειας χρήσης του οδικού δικτύου, μολονότι βέβαια η προσέγγιση αυτή δεν αντιμετωπίζει με ισότιμο απόλυτα τρόπο τις δύο αρχές, ο χρήσης πληρώνει και ο ρηπαίνων πληρώνει. Υπάρχουν βέβαια κάποια εκκρεμή ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο στο οποίο αναφερόμαστε. Αναφερόμαστε σε ένα σφαιρικό πλήρε οδικό δίκτυο Πού ακριβώ όμω από νομική πλευρά θα αρχίσουν να ισχύουν όλα αυτά τα νέα καθεστώτα τα οποία προτείνει η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει επίση να δούμε αν υπάρχουν κάποιες άλλες συναλλακτικέ λύσεις, ορισμένα κράτη-μέλη, και αν μπορούν αυτά να αποφασίσουν σε ποιε περιφέρειές του θα μπορούν να επιβάλλουν συγκεκριμένου κανόνε στα ΙΟΤΑΧΗ. Θεωρούμε εμεί ότι τα ΙΟΤΑΧΗ αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία. Και αυτό διότι είναι επιβατικά αυτοκίνητα, και ουσιαστικά δεν ασχολούνται με οδικές διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και δεν ε, εμπλέκονται καθόλου στον ε, εμπορικό οικονομικό ανταγωνισμό. Οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί το γιο ταχύ του. Θα θέλαμε λοιπόν κάπου στη νομική βάση της νέας αυτής πρότασης ε, να υπάρχει μία βάση τελικά δεδομένων που ουσιαστικά να δείχνει στα κράτη-μέλη τι κάνουμε με τα χρήματα εκείνα τα οποία συλλέγουμε από τους αυτοκινητοδρόμους και πώς αυτά επανεπενδύονται στη συνέχεια προκειμένου να παράσχουμε υπηρεσίες υψής της ποιότητας στους δρόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, μία ακόμα πρόταση είναι η απόφαση για το EETS Πώς μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε σε σχέση με την οδική τιμολόγηση. λέγεται λοιπόν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούν όλα αυτά να επιτευχθούν μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων, EETS. Υπάρχουν πολλά στοιχεία εδώ πέρα τα οποία πρέπει να προασπίσουμε. Σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα διοδίων μπορούν όντως να λειτουργήσουν στην πράξη. υπάρχει τουλάχιστον ένα ηλεκτρονικό σύστημα τηλεδιοδίων σε κάθε κράτος μέλος το οποίο να λειτουργεί στην πράξη. Αυτή τη στιγμή στο εξασφαλίσουμε αυτό θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο. Βάσει λοιπόν της εθνικής πραγματικότητας περνάμε στο περιφερειακό επίπεδο και εφόσον όλα λειτουργούν σωστά και έχει οριμάσει η αγορά και υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι παράγοντες στην αγορά, τότε μόνο μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα τηλεδιοδίων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων θα πρέπει όμως να θεωρείται ότι είναι ένα είδος αγοράς. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμεί κανόνες αγοράς, θα πρέπει να ρυθμίζονται με τον φυσιολογικό τρόπο με τον οποίο τελικά εξελίσσονται. Η αγορά ποια ακριβώς είναι, η αυτοκινητόδρομοι τελικά και η πάροχη υπηρεσιών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στους χρήστες των, στο, στις των αυτοκινητοδρόμων και οι οποίοι απαιτούν από αυτούς την καταβολή τελών. Ξέρετε ότι δεν είναι καλόβουλοι όλοι οι χρήστες, δεν πληρώνουν όλοι αγόγγιστα τα διόδια τους, τα οδικά τους τέλη. Είτε ακούσια είτε ακούσια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς επιβολής της νομοθεσίας έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι ένας χρήστης που χρησιμοποιεί ένα δικό δίκτυο όντως καταβάλει τα τέλη που τον αναλογούν. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε διασφαλίσει. Πρέπει να καταφέρουμε να εντοπίσουμε και να διευκρινίσουμε ακόμα κάποια κρεμή προβληματικά ζητήματα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια θέματα τα οποία πρέπει να διευθετήσουμε. Εμείς διαχειριζόμενοι πολλές φορές τους αυτοκινητόδρομους και το δικό δίκτυο, δεν γνωρίζουμε καλά πώς έχουν τα πράγματα σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα συστήματα ισχύουν στην Νότια Ιταλία, Άλλα συστήματα οδική τιμολόγηση έχουμε στη Βόρεια Γαλλία, για παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα, έτσι ώστε κάθε πολίτης κάθε μπλεκόμενος παράγοντας να μπορεί πραγματικά να γνωρίζει τι συμβαίνει σε κάθε τμήμα του οδικού δικτύου και σε κάθε επιμέρους τμήμα του ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιοδίων. Γι' αυτό το λόγο πραγματικά θέλουμε να γνωρίζουμε αφενός μεν τι έχει συμβεί στο παρελθόν και πώς αποτιμά τη χρήση του, για παράδειγμα η Ευρωβινιέτα, και θα πρέπει επίσης να δούμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ποιοι κανόνες θα ισχύσουν και πώς οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται στην πράξη, ποιος θα παρακολουθεί τελικά την αποτελεσματική εφαρμογή του. Σας ευχαριστώ κύριε Διονέλη. Έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη παρουσίαση των ε, προσκεκλημένων μας. Ευχαριστώ όλους που ήταν πειθαρχημένοι χρονικά. Ελπίζω και τα μέλη να είναι εξίσου πειθαρχημένα. Τα μέλη έχουν μπροστά τους την κατανομή, γνωρίζουν πόσο χρόνο έχουν στη θέση τους. το κάθε μέλος που θέλει να παρέμβει θα θέσει ερωτήσεις και εφόσον η απάντηση λάβει αρκετό χρόνο δεν θα μπορέσει το μέλος να θέσει και άλλη ερώτηση. Θυμίζω. Και παράκληση και πάλι στα μέλη του πάνελ να είναι όσο αποτελεσματική γίνεται στις απαντήσεις προς τα μέλη δεν μπορούμε να πάμε σε μακροσκελείς τοποθετήσεις γιατί ίσως κάποιες ερωτήσεις να ξαναυποβληθούν. Εν πάση περιπτώσει παρακαλώ να αποφύγουμε τις μακροσκελείς τοποθετήσεις για να μπορέσουμε να απαντήσουμε όσο περισσότερες ερωτήσεις γίνονται. Ας είμαστε όλοι παρακαλώ αποτελεσματικοί. Θα ξεκινήσω με την κυρία εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Κριστίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, το αναφέρατε με κάποιο τρόπο, αλλά και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Η βασική αρχή της οδηγίας είναι Αφενός ο ρηπαίνων πληρώνει και αφετέρου ο χρήστης αναλαμβάνει επίσης ένα κόστος. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συνάπιες, συνέπειες που απορρέουν από τη χρηματοδότηση των ειδικών δικτύων. Υπάρχει μια σημαντική ανησυχία που σχετίζεται με τη ρήπανση. Αναφέρθηκε από τους ομίλητες, αλλά προς την κυρία Κρή, σχετικά με την, τις υποδομές που βρίσκονται σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση και καθότι έχουμε και τελείως διαφορετικά συστήματα μεταξύ της μίας και της άλλης χώρας θα έπρεπε να, εναρμονίσ... να εναρμονίσουμε κάπως τα συστήματα αυτά και να μην μείνουμε στην κατάσταση που έχουμε σήμερα. Θεωρείται λοιπόν ότι αν είχαμε μία σύνδεση των ε, κονδυλίων κατά τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαν να, έχουν, να μειωθεί ο αριθμός ε, των χρηστών που θα υπόκεινταν στα τέλη αυτά. Κυρία Κρίντ, κοιτάξτε αυτό το earmarking που, στο οποίο αναφέρεστε. Ε, στην ουσία ε, είναι μία από τις μεθόδους που έχουμε σχετικά με τα κονδύλια που θα δεσμευθούν από τους προϋπολογισμούς. Αλλά Νομίζω ότι μάλλον κατευθύνεστε προ τελικώ τον προπολογισμό των κρατών μελών, από ό,τι καταλαβαίνω. Προς τον κύριο Λεμπεντά τώρα τη IRU, επιθυμείτε να υπάρξει μια, διαφορο... μια διαφορετική μεταχείριση για τα λεωφορεία, μια εξαίρεση. Δεν πιστεύετε αν επανέλθουμε στις βασικές αρχές ρηπαίνων πληρώνει και χρήστης πληρώνει, το πιο αποδεκτό θα ήταν όλα τα οχήματα να τα αφορά η υποχρέωση ανάλογα όμως με το ποσοστό ρήπανσης του κάθε οχήματος και αυτή η αρχή να εφαρμόζεται σε όλα ανεξαρτήτως τα οχήματα που ισχύει σε κάποιες χώρες σήμερα αλλά δεν έχει εναρμονιστεί. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, πρόκειται για ερώτηση που αφορά στην πολιτική βούληση είχαμε την πολύ πρόσφατη πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση των κανόνων αγοράς ε, για τα πούλμαν και τα λεωφορεία. Εάν αυξήσουμε το ποσοστό της ε, αγοράς, της συμμετοχής τους, έχουμε θετικές επιπτώσεις ως προς το περιβάλλον, ως προς την, ε, την κοινωνική διάσταση. Όχι, δεν ήταν αυτή η ερώτησή μου, κύριε. θα ήθελα να απαντήσετε στην ερώτησή μου. Δηλαδή, δεν θα ήταν πιο σωστό, πιο δίκαιο το σύστημα αν τα τέλη επιβάρυναν όλα τα οχήματα ανάλογα με το ποσοστό ρηπάνσεών τους, διότι η οδηγία προβλέπει για τις δύο αρχές, όπως έλεγα, ρηπαίνων και χρήστης. Επομένως, ανάλογα με το είδος της μετακίνησης, το είδος της χρήσης του συγκεκριμένου οχήματος, δεν νομίζετε ότι θα ήταν μια αρχή σωστή. Κοιτάξτε, ε, ως προς το κόστος του δικτύου ναι, αλλά ως προς το εξωτερικό κόστος η απάντηση μου είναι όχι. Πρέπει να είμαστε ευνοϊκοί προς το είδος αυτός ε, μεταφορών για το εξωτερικό κόστος. Ε, κοιτάξτε, το εξωτερικό κόστος σχετίζεται με τη ρήπανση. Τα πούλμαν σήμερα δεν είναι καθαρά οχήματα, θα το αναγνωρίζετε φαντάζομαι αυτό. Ζητάτε λοιπόν μία εξαίρεση χωρίς να αναγνωρίζετε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, πρέπει να λάβει κανείς ε, τον αριθμό των επιβατών που μετακινούνται με κάθε όχημα για να υπολογίσουμε πόσο, πόσο ρηπογόνα είναι. Η πιο βιώσιμη μέθοδος μεταφορών για τους Ευρωπαίους πολίτες σήμερα είναι τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Σας ευχαριστώ, διακόπτει ο Πρόεδρος. Και θα πάμε τώρα στο δεύτερο εισηγητή, ο κύριος ο κύριο Σαλίνη, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω προς τον κύριο Μπενεντέτο και προς τον κύριο Διονέλη. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που μας λέτε ότι τα τεχνολογικά πρότυπα όσον αφορά τα τηλεδιώδια δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προβλέπονται σε ένα παράρτημα. Νομίζω ότι επ' αυτού ουσιαστικά πρέπει να συμφωνεί το Συμβούλιο και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τεχνικής πλευράς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην ε, συχνότητα που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα συστήματα τηλεδιοδίων και τα συστήματα εφιούς ε, οδήγησης. Μάλιστα, μια αντιπροσωπεία από τις Πολιτείες για τις μεταφορές είχε ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Η Επιτροπή προτείνει, προτείνει η συχνότητα για τα τηλεδιόδια να περάσει στα 5,9 GHz, που είναι η συχνότητα που χρησιμοποιούν και τα συστήματα εφιούς οδήγησης. Θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα οδηγήσει σε περιττέρω δαπάνη ή θεωρείτε ότι μπορούν να συνεπάρχουν δύο διαφορετικές συχνότητες 5,8 και 5,9 GHz. Λοιπόν, για ποιο λόγο πρέπει να περάσουμε στο νέο αυτό σύστημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το σύστημα με τα 5,8 GHz. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε αυτή τη στιγμή σε μια άλλη συχνότητα, αλλά εδώ πέρα νομίζω το κόστος για την υιοθέτηση της νέας αυτής τεχνολογίας θα είναι υψηλό. Από τεχνολογικής πλευράς, απευθύνομαι στον κύριο Σαλίνη, το να έχουμε παράλληλα δύο συχνότητες μπορεί πραγματικά να προκαλέσει παρεμβολές η μία στην άλλη και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι αρκετά σαφές, αρκετά συγκεκριμένο. Επομένως, η υπόθεση ήταν να διατηρήσουμε τη συνύπαρξη των δύο αυτών συγνωτήτων. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο να σταματήσουμε την εφαρμογή των συστημάτων εφιούς οδήγησης. Εσείς θεωρείτε αυτή τη στιγμή ότι έχει οριμάσει αρκετά η χρησιμοποίηση της συχνότητας 5,8 στα τηλεδιώδια ή θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει έπειτα η χρήση της συχνότητας 5,9 να χρησιμοποιηθεί αυτή δηλαδή σε ευρύτερο επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο σας ρώτησα κιόλας αν σε κάποια φάση στο μέλλον μπορούν να συνεπάρξουν οι δύο αυτές συχνότητες. Ε, Θεωρούμε λοιπόν ότι μπορούν οι δύο αυτές τεχνολογικές επιλογές να συνεπάρξουν ή ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η μετάβαση σε μία και μοναδική συχνότητα στο μέλλον. Ή θεωρείτε ότι και στο μέλλον μπορούν οι δύο συχνότητες να συνεπάρξουν. Απάντηση. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολη και δαπανηρή η συνύπαρξη των δύο συχνοτήτων των δύο συστημάτων. Είναι πολύ πολύπλοκο και ιδιαίτερα δαπανηρό να υπάρχουν παράλληλα δύο συχνότητες και μάλιστα υπό το φω, μάλιστα αυτού το οποίο λέγατε ότι θα έχουμε όλο και περισσότερα οχήματα τα οποία θα λαμβάνουν μηνύματα από τους δορυφόρους ε, όλα αυτά τα αυτοοδηγούμενα οχήματα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να περάσουμε από τη συχνότητα 5-8 σε μια λύση που θα είναι καθαρά δορυφορική. Να απευθυνθώ και στον κύριο Διονέλη. συμφωνείτε την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο άρθρο 6 όπου αναφέρεται στο enforcement στην επιβολή δηλαδή της νομοθεσίας και στο όλο το σύστημα της παρακολούθησης του follow-up. Ποιος όμως θα πρέπει να ασχοληθεί με τα συστήματα αυτά follow-up. Δεν είναι αυτό σαφές ακόμα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θεωρείτε ότι αυτό για τους ανθρώπους που εσείς εκπροσωπείτε θα μπορούσε να οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλέ δαπάνες. Πολύ σύντομα, λέει ο πρόεδρος, πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Το ζήτημα της επιβολής της νομοθεσίας και του ελέγχου της εφαρμογής θα μπορούσαμε πάντα να λέμε το ίδιο πράγμα, ότι τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά στον τομέα των διοδίων αν δεν υπάρχει το enforcement, η επιβολή της νομοθεσίας. Τρεις είναι εδώ πέρα βασικά. Ο χρήστης καταρχάς, αυτός που χρησιμοποιεί τελικά την υποδομή, αλλά ο χρήστης αυτός δεν έχει μία σύμβαση με, τον, με την υποδομή των διοδίων, αλλά με τον πάροχο της υπηρεσίας. Άρα μιλάμε για ένα τρίγωνο, μια τριγωνική σχέση, η οποία κάπως θα πρέπει να υπάγεται σε ένα σύστημα παρακολούθησης και εφαρμογής νομοθεσίας. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια επιβολή της νομοθεσίας τη στιγμή που εμπλέκονται τρεις παίκτες, τρεις παράγοντες, όπως σας είπα. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Πρέπει όμω αυτή τη στιγμή να συντομεύουμε. Δεν μπορούμε να υπερβαίνουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον χρόνο αγόρευση. Διαφορετικά θα καταφέρω να πάρω το λόγο και οι υπόλοιποι ομιλητέ. Η κυρία Κλούν τώρα μπορεί να πάρει το λόγο, που είναι και αυτή η συγγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Τότση σε ό,τι αφορά το earmarking των ε, τελών για τη χρήση του δρόμου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα να μου απαντήσει ο κύριος Τόρτς από το D&D. Ως γενικό κανόνα δεν θεωρούμε ότι το earmarking αποτελεί καλή ιδέα. Πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίσουν πώς θα δαπανούν τα χρήματα αυτά, τα έσοδα αυτά και ενδεχομένω να χρειάζεται χρήματα σε σχολεία, σε νοσοκομεία και όχι στους δρόμους. Δεν νομίζουμε ότι βγάζει νόημα το earmarking. Ευχαριστώ. Εξαιρούνται τα λεωφορεία από, τις, τα σχετικά τέλη. Έχει νόημα αυτό. Συμφωνώ ότι τα πούλμα και τα ελεοφορία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο όλο σύστημα των μεταφορών, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε προ ένα σύστημα όπου όλα τα οχήματα θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμολόγηση αυτή τη χιλιομετρική. Και φυσικά αυτό περιλαμβάνει και τα πούλμα. Και προ τον κύριο Λίπερ, μια ερώτηση. Το κόστο για το HIV. Είπατε ότι 130% ε, καλύπτουν του κόστου ε, συντήρηση των δρόμων. Τι πιστεύετε για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση της φορολογίας σε ό,τι αφορά και το συνδυασμό με το κόστος ε, συμφόρησης. Ναι, κοιτάξτε, εφόσον ε, θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ιδιαιτερότητα των εσόδων, την ίση δηλαδή, το ίσο επίπεδο εσόδων, ε, ναι, φυσικά. Να ρωτήσω και για τα οχήματα χαμηλού κόστους ε, που θα συμπεριληφθούν και αυτά. Έχετε κάποια πρόταση και τι θα γίνει σε ό,τι αφορά το διασυνοριακό επίπεδο. Ιδιαίτερως ε, στην κεντρική Ευρώπη όπου χρειάζεται κανείς να περνάει πολλά σύνορα θα περιοριστεί κάπως η απόσταση. Έχετε κάποια άποψη και έχετε σκεφτεί το θέμα των ε, οχημάτων χαμηλού κόστους, γιατί βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται όντω περισσότερο αυτά τα οχήματα. Εννοείται τα ελαφριά οχήματα. Ναι, κοιτάξτε, αν ε, μπορούμε να δείξουμε ότι η χρήση τέτοιων οχημάτων, ελαφριών οχημάτων ε, για τις δεσμευτικές μεταφορές φτάνει σε ανησυχητικά επίπεδα, θα πρέπει να υπάρξει κάποιο νομοθεσία, κάποια ρύθμιση τώρα κατά πόσο αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να συμβάλλουν στο πλαίσιο του, της Ευρωβινιέτας ε, και πάλι αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε είναι τι, πόσο συνεισφέρουν στο κόστος σήμερα και κατά πόσο μας ικανοποιεί το επίπεδο αυτό. Και κύριε Τόντ, πείτε μας για τα ελαφριά οχήματα. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο να εξαιρεθούν μέσα στα σύνορα μια χώρας και όχι στις διασυνοριακές μεταφορές. Πρέπει να σας πω ότι για μένα το θέμα των διασυνοριακών μεταφορών δεν έχει να κάνει τόσο πολύ, δεν είναι τόσο σχετικό. Έχουμε διάφορες ευρωπαϊκές νομοθεσίες που προωθούν τα ελαφριά οχήματα. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο λοιπόν μεροληπτεί. Και νομίζω ότι το δίκαιο θα ήταν να γίνουν αλλαγέ στην νομοθεσία, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, προκειμένου να πετύχουμε πάλι ισορροπία μεταξύ των οχημάτων αυτών. Και μία ερώτηση για τον κύριο Λόχμαν, αν μου επιτρέπετε. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρξει τιμολόγηση χιλιόμετρακή ε, σε όλους τους ε, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις αποστάσεις. Αυτό δεν θα ήταν διακριτική μεταχείριση κατά των μικρών χωρών και κατά των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί και πάλι αν το συγκρίνουμε με τους ε, έχουμε και πάλι χώρες με μικρό σιδηροδρομικό δίκτυο και το τέλος, τα τέλη αφορούν όλη την απόσταση και το τελευταίο χιλιόμετρο. Άρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει οικονομικός αντικτύπωση. Σας ευχαριστώ. Ακριβώς έτσι πρέπει να κάνουμε. Να θέτουμε ερωτήσεις και να έχουμε γρήγορες απαντήσεις. Ε, ευχαριστώ αυτόν που απήντησε ε, για τον τρόπο με τον οποίο απήντησε γιατί δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Βάντερ Κάμπ, τρία λεπτά. Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Σας ευχαριστώ. Όχι, μία ερώτηση έχω να κάνω σε δύο άτομα καλύτερα. Πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Πενιτέτο. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς θέλετε. Θέλετε ένα σύστημα για διάφορες επιχειρήσεις ή θέλετε διάφορες συστήματα για διαφορετικέ επιχειρήσει. Και το, κύριο, το ίδιο ερώτημα απευθύνω και στον κύριο Διονέλη. Ένα σύστημα για διάφορε εταιρείε ή διαφορετικά συστήματα για διαφορετικέ εταιρείε. Io penso che la standardizzazione Κοιτάξτε, εγώ θα προτιμούσα ένα σύστημα ή στα πλαίσια του οποίου διάφοροι φορείς θα μπορούσαν να ανταγωνίζονται ισότιμα. One is okay, but has to be Ένα σύστημα που πρέπει να είναι λειτουργικό. Πολλά σύστημα πρέπει να είναι διαλειτουργικά και αυτό είναι πιο δύσκολο. Μάλιστα και μία ερώτηση προς τον κύριο Μπενιντέτο. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των διοδίων και των έξυπνων ταχογράφων. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα κανένας άμεσος σχετισμός. Ίσως στο μέλλον να υπάρξει μια σύγκληση μεταξύ ταχυγράφ και διοδίων. Ίσως όχι τόσο για τα διόδια καθεαυτά, αλλά για την προστέμενη αξία που θα μπορούσε να δίνει αυτό στον ε, μεταφορέα. κύριε Τότσα, στο Συμβούλιο φαίνεται ότι γίνεται μια συζήτηση μεταξύ του θέματος της επικυριαρχίας και αυτών που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα σύστημα, αλλά τα κράτη, για παράδειγμα, τα, για τα γιοταχή στην Ολλανδία να μπορούν να αναστείλουν το σύστημα αυτό. Νομίζω ότι η συζήτηση για την επικυριαρχία δεν είναι και τόσο δύσκολη. Νομίζω ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθούν διαφορετικά συστήματα, βινιέτε. Μάλλον οι βινιέτε και τα διαφορετικά συστήματα θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά. Δεν έχουν και θέση στην κοινή, αγορά. Και τώρα, αν θέλουν τα κρατημέλη να επιβάλλουν α, οδικές ε, οδική χρέωση μπορούν να επιλέξουν να το κάνουν αυτό, χιλιομετρική για παράδειγμα τιμολόγηση, ή να μην το κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κύριο Κάμπ, λέει ο πρόεδρο, και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Έρτουγ για δύο λεπτά. Καλημέρα σα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω το εξή. Το 75% περικοπή για τη χρήση των δρόμων είναι καλό και θα πρέπει να ευτερηθεί. Και εγώ πιστεύω ότι το Ήρμαρ και η Κυριτότσα έχει νόημα. Καλό θα ήταν ε, αν όλε οι κυβερνήσει βάζουν τα λεφτά του και τα επένδυαν σε σχολεία και νοσοκομεία. Ε, δεν το κάνουν όμω, γι' αυτό έχει νόημα το earmarking, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό ε, να χρήματα αυτά να μην πηγαίνουν σε εξοπλισμού. Αυτό είναι όμω πολιτικό ζήτημα. Μία ερώτηση. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι μας λείπει μία σύγκριση της επιβάρυνσης κόστους των διαφορών τρόπων. Αυτό εξακολουθεί να λείπει και αυτό εκφράζεται και στις παρεμβάσεις. Αυτό που σημείωσα και σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να κοιτάξω γιατί δεν έχω και παραπάνω χρόνο. Ο κ. Λεπέντε λέει από το αεριού ότι τα ευρωπαϊκά φορτηγά καλύπτουν 130% του κόστους τους και στη συνέχεια ο κύριος Λόχμαν αναφέρει ότι μόνο το 30% του κόστους ε, καλύπτεται. Μα ποιο από τα δύο αληθεύει τελικά. Δεν έχω και πολύ χρόνο, σας παρακαλώ γρήγορα. Βιαστείτε. Νομίζω ότι το σημείο αναφορά είναι διαφορετικό. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι το δικό μα σημείο αναφορά είναι το τρίτο πλαίσιο Ευρωπαϊκή βινιέτα που καλύπτεται από το τρέχον πλαίσιο δηλαδή και το εξωτερικό κόστο που καλύπτεται ε, από το τρέχον πλαίσιο. Δεν υπερβαίνουμε. Ναι, η βάση είναι διαφορετική, αλλά ο κύριος Τότς θα ήθελε να απαντήσει ίσως εν συντομία. Νομίζω ότι αξίζει να το κοιτάξουμε αυτό πιο εντελεχώς, να κοιτάξουμε τις εκθέσεις και του FIA και του IRU, γιατί εκεί θα δείτε ότι στη μεθοδολογία του έχουν κάνει διάφορες επιλογές, οι οποίες προφανώς επηρεάζουν πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Καθίστε και κοιτάξτε τα λοιπόν. Μάλιστα λοιπόν, θα είχε νόημα να εναρμονιστεί και η μέθοδος της εξαγωγή των ερευνών. Αυτό είναι καθήκον, φαντάζομαι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Η κυρία Φώστερ για τρία λεπτά, τρισήμιση λεπτά. Um, thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, προς τον κύριο Τόντ, δεν θα συμφωνούσατε ότι είναι απολύτως λογικό αν θέλουμε να εξωθήσουμε τους ανθρώπους προς άλλα μεταφορικά στήματα από τα αυτοκίνητα, να τους κατευθύνουμε προς τα πούλμαν, π.χ. Γιατί τα λεωφορεία και τα πούλμαν μεταφέρουν πολλούς ανθρώπους, θα μου φαίνεται τελείως παράλογο να τα επιβαρύνουμε κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα γιοταχή. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα το σχόλιο σας επ' αυτού. Γιατί θέλουμε να αυξήσουμε τις λύσεις των δημοσίων μεταφορών. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ευρύτερο πεδίο. Καταρχάς έχουμε μια πρόταση περαιτέρω απελευθέρωσης που θα διευκολύνει την διάβαση των λεωφορείων διαμέσου της Ευρώπης. Επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο τελών να το καταβάλουν. Επομένως ο συνδυασμός είναι λογικός. Ναι, αλλά τότε τι θα έχουμε. Αν επιβαρύνουμε τα φορτηγά, αυτό θα το περάσουν στους επιβάτες. Και στις δημόσιες μεταφορές, μαζικές μεταφορές, ε, προσπαθούμε το κόστος μεταφοράς να το διατηρήσουμε χαμηλό. Ιδιαίτερα για τους πολύ μικρούς και πολύ μεγάλους. Αυτό θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε από αυτού. Αλλά προχωρώ στον κύριο Λόχμαν. Εγώ είμαι παδός των σιδηροδρόμων, νομίζω ότι όλοι είμαστε. Αλλά γιατί είστε τόσο εχθρικοί προς τους ε, φορείς ε, των ε, πούλμαν των οδικών μεταφορών. Όλοι εξαρτώμαστε σε κάποιο βαθμό από αυτούς. Δεν μπορούμε να έχουμε συνδέσεις συνδεδρομικές σε όλο το έδαφος. Και σε κάθε περίπτωση οι σιδηρόδρομοι συνήθως ενισχύονται από τον φορολογούμενο, ενώ οι εταιρείε Πούλμαν ε, όχι. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε, ε, μάλιστα αν επιβαρύνουμε και τους μεταφορείς των φορτηγών, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε υπερβολικά υψηλό κόστος μεταφορών αγαθών. Θα ήθελα επ' αυτόν λοιπόν να σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, μιλώντας για επιδοτήσεις, τι, οι επιδοτήσεις στις υποδομές τι είναι. Κάτι λέγεται εκτός μικροφώνου. Ε, στο συγγνώμη, στο συγγνώμη. Ε, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του πώς λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι και μια εταιρεία που έχει κάποια φορτηγά ή κάποια πούλμαν. Ε, εσείς θέλετε ε, με πάση θυσία να εξασφαλίσετε ότι αυτοί θα επιβαρυνθούν. Ναι, αλλά εδώ ε, προσπαθούμε να διακρίνουμε την επένδυση των υποδομών που ισχύει για το δικό δίκτυο και τους σιδηροδρόμους και της εμπορικής δραστηριότητα που γίνεται υπό διαφορετικές συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία επιδότηση για τους σιδηροδρόμους υπό την έννοια της κυκλοφορίας. πρέπει για να έχουμε συγκρίσιμες συνθήκες να, δούμε και το κόστος που επιβαρύνει τους ε, διερχόμενους από το οδικό δίκτυο για να έχουμε αντίστοιχο κόστος στην πραγματικότητα οι εταιρείε ε, μεταφορών σιδηροδρόμων αυτοί, αυτές επιβαρύνονται διότι αναλαμβάνουν έμεσα το κόστος που επιβαρύνει τις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ τον κύριο Λόχμαν, λέει ο πρόεδρος. Τώρα, 3,5 λεπτά, σε μένα τον ίδιο. Η πρώτη ερώτηση για τον κύριο Τόντς. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, να εντοπίσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε την εξωτερική διάσταση του κόσμου και συγκεκριμένα τη συμφόρηση και την ηχορύπανση. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί όντως αυτό να πετύχει, την εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι εφικτό. Ναι, αλλά δεν ξέρετε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα. Προς τον κύριο Λεμπέντε η επόμενη ερώτηση. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε να έχουμε στα πλαίσια της πρότασης της Ευρωβινιέτας αύξηση των τελών. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε η αύξηση αυτή των τελών να μειώσει το περιθώριο των επιχειρήσεων. Πώς μπορεί να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Απάντηση. Κοιτάξτε. Οι τελευταίες αναθεωρήσεις της Ευρωβινιέτας δείξαν ότι όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, το κόστος μετακυλείται τελικά στον τελικό χρήστη. Στους απλούς πολίτες, σαν και εμένα και σαν εσάς. αν δεν υπάρχει ένας πραγματικός συνταγωνισμό ε, μεταξύ των διαφορετικών μέσων μεταφοράς και τρόπων μεταφοράς, ε, δεν νομίζω τελικά ότι μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Μας λέτε λοιπόν ότι δεν επηρεάζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά επιβαρύνει τελικά τον τελικό καταναλωτή, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να το αναλάβουν το κόστος αυτό, το κάνουν. Διαφορετικά βέβαια οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ενδεχομένως ε, να ζημιωθούν οικονομικά. Τώρα ο κύριος Διονέλης και ο κύριος Μπενεντέτο μπορούν να απαντήσουν στην επόμενη ερώτηση. Θα ήσασταν υπέρ της διαλειτουργικότητας και της απλούστευσης του συστήματος ή προτιμάτε το σύστημα να ανοίξει στον ανταγωνισμό περισσότερο ή πιστεύετε ότι είναι συμβατά και τα δύο, και οι δύο αυτές προσεγγίσεις δηλαδή και αν ναι, Απάντηση. Ναι, οι δύο προσεγγίσεις είναι συμβατές. Μπορούμε να έχουμε διαλειτουργικά συστήματα σε καθεστώς ανοιχτού ανταγωνισμού, ακριβώ αυτό θέλουμε να δούμε. Από την άλλη όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι χρειαζόμαστε εδώ πέρα δύο παράγοντες, τους αυτοκινητοδρόμους και τους παρόχους υπηρεσιών. Εκεί έγκυται η δυσκολία. ο κύριος Μπενεντέτο. Συμφωνώ απόλυτα. Προφανώς οι δύο προσεγγίσεις είναι συμβατές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες στο παιχνίδι, υπάροχοι υπηρεσιών, υπεύθυνοι υποδομής διοδίων και καθεξής. Θα πρέπει ο καθένας λοιπόν να έχει συγκεκριμένε αρμοδιότητες και καθήκοντα. Πρόεδρος και η σχέση ανάμεσα στους, στις αρχές που είναι υπεύθυνε για τις υποδομές και στις αρχές εκείνες που είναι υπεύθυνε για την ίσπραξη της Ευρωβινιέτες. Κύριε Μπενεντέτο, τι έχετε να πείτε προς αυτό. Κοιτάξτε, ως πάροχος υπηρεσιών προφανώς μας ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό. Πρέπει λοιπόν να δούμε εμείς πώς γίνεται η ίσπραξη των τελών και πρέπει να δούμε επίσης αν ο τελικός χρήστης μπορεί πραγματικά να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα καταβάλει τα οδικά αυτά τέλη. Η κυρία Κίλωνεν τώρα έχει το λόγο για τρία λεπτά. Δεν είναι στην αίθουσα, ενδεχομένω να μιλήσει αργότερα. Ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο τώρα για τρία λεπτά. Μία ερώτηση προς τη Λεβέντα. Αν ε, συμπεριληφθούν οι Βρυξέλλες, ε, αν εξαιρεθούν οι Βρυξέλλες από τα τα διόδια. Συμφωνείτε να υπάρχουν, να απαλλαγούν και τα διόδια οι συνδρομικές γραμμές. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πέρα από την φορολόγηση των υποδομών. Έχει να κάνει με το συνολικό πλαίσιο φορολόγηση για όλα αυτά τα ζητήματα για να λεφτούν τέτοιε αποφάσει. Μια ερώτηση προ την κυρία Κρέιτ. Στη Γερμανία 53 εκατομμύρια συλλέγονται από του φόρου και από τα διόδια και αυτά τα έσοδα που ιστορικοποιούνται είναι 20 εκατομμύρια κάθε, χρόνια, χρόνο. Πώς καταλήγεται στα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε η έρευνα έγινε από το συντέλευτη και δεν περιλαμβάνει το εξωτερικό κόστος γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αβεβαιότητα για το πώς υπολογίζονται που δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Μία ερώτηση προς τον κύριο ε, το ίδιο ρύθμιση για όλους για τα ηλεκτρονικά για τα, για ηλεκτρικά ε, οχήματα χωρίς ε, απαλλαγές ε, και για, τους και για τα ηλεκτρικά τρένα. Θα ήταν καλό το παράδειγμα που θα οδηγούσε στον σωστό ανταγωνισμό. Νομίζω ότι ό,τι αφορά τις δικές μεταφορές έχουμε πρόβλημα με τις εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα, να δώσουμε ένα ενιαίο μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την αγορά, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εταιρείε να επενδύουν. Και μόλις καταφέρουμε να υπάρχει ένα μερίδιο σωστό τέτοιων οχημάτων, να καταργήσουμε αυτά τα κίνητρα. Ερώτηση προς τον κύριο Λόχμαν, earmarking, αν ισχύσει μόνο για τις ε, οδικές μεταφορές, θα βοηθούσε αυτό την μετάβαση στους δρόμους, ότι την επιτάχυνε, το οποίο και αποτελεί γενικότερη άρχη, ή μήπως θα την παρεμπόδισε είσαστε και επίσης υπέρ του earmarking για τους των οδικών μεταφορών όπως γίνονταν στην Ελβετία. Μόνο για το σύστημα διοδίων, όχι σε ό,τι αφορά το earmarking για, το, για την αρχή του ορυπαίνου πληρώνει. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Λιμπιντάκη και στην κυρία Κρήτη Στην Ισπανία τα ευρωπαϊκά χρήματα δαπανούνται για την ε, κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και στα αυτοκινητοδρόμους υπάρχουν ε, διόδια και στις εθνικές ε, γίνεται μεγάλη γίνεται συμφόρηση. Θα ήσασταν υπέρ του να ισχύσουν σύστημα διοδίων για όλους τους δρόμους, για όλα τα δικά δικτύα, για να μην υπάρχει μεταφορά σε μικρές αρτηρίες. Κοιτάξτε, Υπάρχει όντως ε, κίνδυνος μετάβασης ε, της κυκλοφορίας σε μικρές αρτηρίες. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η επιρροή των διοδίων αυτών στους ε, πολίτες δεν συγκρίνεται και θα μπορούσε να επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση πολλών οδηγών που δεν έχουν άλλες επιλογές. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λούγκριν. Όχι, ζητώ συγγνώμη κυρία Σίμερ. Τρία λεπτά παρακαλώ κυρία μου. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Περισσότερο δήλωση παρά ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι άλλα συστήματα χωρών για τα τέλη, για τα οδικά τέλη είναι αποδεκτά. Εμείς το είχαμε απορρίψει. Και είχαμε και προτάσεις με μαζική στήριξη, 2 εκατομμύρια υπογραφές κατά των διοδίων. Εμείς δεν επιθυμούμε λοιπόν ε, τα συστήματα διομοίων. Ήδη οι οδηγοί θεωρούν ότι πληρώνουν, καταβάλουν υπερβολικό κόστος. Υπάρχει και το σχετικό κόστος ε, για τα οργανωτικά. Οι εταιρείε κατασκευής των οδικών δικτύων ε, υφίστανται τεράστια πίεση για πιο καθαρά συστήματα, αλλά οι οδηγοί τελικώς επιβαρύνονται συνεχώς, βλέπουμε και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν όλο και πιο καθαρά ε, μικρά φορτηγά, ε, πιο καθαρά δηλαδή για, τα, για τις μεταφορές του μέλλοντος, αλλά αυτά δεν είναι ακόμα διαθέσιμα. Γιατί λοιπόν επιβαρύνουμε με όλη αυτή την πίεση τους τελικούς χρήστες, τους οδηγούς τα, τα διόδια τελικώς χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση των οδικών δικτύων και τίποτε άλλο. Στο Ηρωμένο Βασίλειο τα έχουμε απορρίψει επανειλημμένω και δεν θεωρώ ότι οι προτάσεις οι σημερινέ δεν έχουν κανενός είδου λογική είτε για τους οδηγού μας είτε για τους μεταφορεί μα, οι οποίοι στο τέλος θα πληρώνουν και περισσότερα. Έχετε ερωτήσει για το πανέλ, λέει ο πρόεδρο κυρία Σίμορ. Ε, όπως είπα, πρόεδρε, ήταν δήλωση και όχι τόσο ερώτηση. Γιατί απλώς λέω ότι αυτές οι ιδέες δεν αφορούν στην Βρετανία. Μάλιστα. Η κυρία Άχνου του για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Προς τον ε, κύριο Λεμπεντά και την κυρία Κρίντ σας άκουσα πολλέ φορέ να αναφέρεστε και σωστά στην αρχή της επικροικότητα. Ο κ. Λεμπεντά έκανε ένα πολύ θετικό σχόλιο λέγοντα ότι το βασικό θέμα είναι να καταλάβουμε πού κατευθύνονται τα έσοδα, τα δημόσια κονδύλια. Πού κατευθύνονται δηλαδή αυτά που επιβαρύνουν το φορολογούμενο. Είχαμε το, το ευρωπαϊκό τέλος κυκλοφορίας που αρχικά υποτίθεται ότι θα υποστήριζε τους ανθρώπους με αναπηρία, τελικά εξετράπη. Εν πάση δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα φορολόγησης. Ε, κάποιες χώρες λένε ότι οι οδικοί, οι αυτοκινητόδρομοι πρέπει να είναι δωρεάν, άλλοι όχι. Ε, κάποιοι έχουν κάποια τέλη κυκλοφορίας, κάποιοι έχουν κάποια άλλα συστήματα τελών και τα κτλ. Υπάρχουν διάφορα λοιπόν συστήματα χρηματοδότησης. Επομένως κατά την άποψή σας, καθότι τελικώς οδηγούμαστε σε διάφορα μέτρα, για να το πούμε έτσι, επιβαρυντικά για τον πολίτη, φορομπηχτικά. Πώς θέλετε τελικώς λοιπόν να χειριστούμε την, την επιβάρυνση του παρόντος άνισου συστήματος από επιπλέον μέτρα ανισότητος. Η ερώτησή μου είναι προς τον κύριο Λεμπεντά και την κυρία Κρίντ. Ευχαριστώ κυρία μου. Ε, όπως έλεγα στην παρουσίαση προηγουμένως, η αναθεώρηση του, συστήματος του συστήματος Ευρωβινιέτας ο, ο μόνος ισότιμος τρόπος να, να την δει κανείς θα ήταν να διανεμηθεί το έσοδο προς τις ίδιες οδικές μεταφορές ώστε αυτές να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο καθαρές. Να συμπληρώσω για την επικουρικότητα είναι μια πραγματική ερώτηση. Λέει η κυρία θα έχουμε μια πιο λεπτομερή μελέτη την οποία θα σας υποβάλουμε εντός του Δεκεμβρίου Εμεί θεωρούμε ότι η αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διευκολύνει το γεγονό ότι οι επιβάτε, οι πολίτε ε, να μπορούν να διέρχονται μεταξύ των κρατών, διαλειτουργικό λοιπόν πραγματικά σύστημα, να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα. Ε, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δίνει ένα πλαίσιο εντό του οποίου τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν να περάσουν σε μια επιβάρυνση που τη θεωρούν κατάλληλη για το δικό του έδαφο, για τη δική του επικράτεια. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι όντως αυτό είναι το πλαίσιο των προτινόμενων μέτρων. Είναι ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με την καλύτερη εφαρμογή των όσων υφίστανται σε εθνικό επίπεδο. Ναι, ναι, αλλά η Ευρωβινιέτα δεν είναι απλώ νομικό πλαίσιο, είναι κάτι το οποίο υποβάλλεται εκ των άνω, λέει η κυρία Κρήτο. Ο κύριο Μπάχτορ έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση να κάνω προς τον κύριο Λιβιτά. Στις ε, εξηγήσεις σας ε, ζητήσατε πάρα πολλές εξαιρέσεις και μάλιστα ζητήσατε και άλλους, ε, άλλα σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και πώς θα είναι και δίκαιο πώς θα αποτρέψουμε τις διακριτικές μεταχειρήσεις άμα αρχίσουμε πάλι ε, ένα σωρό εξαιρέσεις και απαλλαγές. Νομίζω ότι οι δύο βασικές εξαιρέσεις ε, για τα λεωφορεία και τα πούλμαν και η δεύτερη για το κόστος συμφόρησης, αυτές οι δύο ουσιαστικά ζητήθηκαν. Θα πρέπει να το δούμε αυτό στο σύνολό του, όχι μόνο στη φορολόγηση των μεταφορών, αλλά λάβουμε υπόψη το ΦΠΑ, το κόστος της φορολόγησης των καυσίμων, της φορολόγησης των οχημάτων οι δύο αυτές εξαιρέσεις λοιπόν, οι δύο αυτές απαλλαγές που αναφέρθηκαν, μου φαίνεται ότι όχι μόνο έχουν πολιτικό, πολιτική σκοπιμότητα, για την προώθηση των δημοσίων συγκοινωνιών, αλλά θα μειώσουν και τη συμφόρηση. Άλλη μια ερώτηση προς την κύριε Τότς τώρα. Είπατε ότι ο θόρυβος και η συμφόρηση θα πρέπει να φορολογούνται και ότι αυτό είναι δυνατόν. Πιστεύετε ότι αυτό θα απαλλάξει από το θόρυβο και από τη συμφόρηση ή μήπως απλά θα μετακυλήσουμε το κόστος στους χρήστες, στους πολίτες. Για τον θόρυβο αν δεν υπάρχει κάποια διάκριση, κάποια διαφοροποίηση, ναι, αυτό θα συμβεί. Γιατί ουσιαστικά θα μετακυλιστεί το κόστος σε αυτούς που προκαλούν το θόρυβο. Είναι διαφορετική η περίπτωση αυτή από την διαφοροποίηση Euroclass. Τρίτη ερώτηση προς τον κύριο Δονέλη. Είπατε ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα, ευρωπαϊκό επίπεδο, εθνικό και τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των φορτηγών και, ποιοι, και ποιες αντικές αρτηρίες εννοούνται. Θα μπορούσατε να μας αναλύσετε λίγο παραπάνω αυτό το στοιχείο. Ναι, βεβαίως. Ο βασικός ε, κανόνας είναι η χιλιομετρική χρέωση. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να πληρώνει ο χρήστης και ο Ωστόσο, όταν μιλάμε για την θελευτική φύση των προτάσεων, κατανοούμε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία προτείνουν στις περιφέρειες, επειδή υπάρχουν διάφορες ευαισθησίες, να ε, απαλλάσσονται τα γητοχεία από τη χιλιομετρική χρέωση και να βασίζονται μόνο στην Ευρωβινιέτα. Αυτό είναι μία λύση την οποία αν επιθυμεί να εφαρμόσει το κράτος μέλος μπορεί να την εφαρμόσει αλλά επί της αρχής η χιλιομετρική χρέωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να προωθηθεί η αρχή του ρηπαίνων πληρών και του χρήστης πληρώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σενάλοβα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια ερώτηση για τον κύριο Διονέλη και τον κύριο Μπενεντέτο. σε σχέση με τα όσα είπατε για την περίοδο των 24 μηνών, ότι δεν είναι ρεαλιστική η περίοδος αυτή. Θα ήθελα να γνωρίζω για ποιο λόγο διατείνεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Μπενεντέτο είπε ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τη χρονική αυτή περίοδο των 24 μηνών. Ποια είναι η άποψή σας για την βαθμία εφαρμογή μέσω περιφερειακών πρωτοβουλειών. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση όσον αφορά τη χρονική περίοδο, γιατί σχετίζεται με το πόσες χώρες είναι έτοιμες να αποδεχθούν τους παρόχους ε, υπηρεσιών, τους service providers. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για το business case, για ένα επιχειρηματικό μοντέλο και να δούμε ακριβώ πώ μπορεί να εφαρμοστεί. Ο κύριο Διονέλη, μα οι ίδιε αγορέ έχουν αποδείξει ότι η περίοδο των 24 μηνών δεν είναι ρεαλιστική. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθεί και εκτό από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό το λόγο είπε επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει μια βαθμιαία σταδιακή εφαρμογή. Α δούμε πρώτα τι γίνεται σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο και ας περάσουμε επίτα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δούμε ότι σε 24 μήνες μπορούμε να έχουμε παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι να μπορούν να λειτουργούν και στην Ιρλανδία και στην Κρήτη για παράδειγμα, τότε ας το κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι η πιο συνετή προσέγγιση είναι να προχωρήσουμε πιο σταδιακά και πιο βαθμιαία. Μία ακόμα ερώτηση. Αναφερθήκατε στη μη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων, ή ETS. Βάσει ποιας εμπειρίας το λέτε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, η ets βασει ποια εμπειρια ιδέα είναι η ολη ιδεα ειναι η εξη Αν συμφωνήσουμε όλοι για τη νέα αυτή πρόταση, θα έχουμε τελικά service providers, παρόχους υπηρεσιών δηλαδή, οι οποίοι θα επεμβαίνουν και θα χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Ακόμα και αν τους ονομάζουμε παρόχους υπηρεσιών ή e ETS, δεν θα καλύπτουν όλη την Ευρώπη, θα καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος, με απότερο στόχο να καλυφθεί όλη η Ευρώπη. Ουσιαστικά θα είναι περιφερειακοί παράγοντες, περιφερειακοί φορείς και όχι ευρωπαϊκοί φορείς εκ πρώτης όψεως αλλά με το να συνεργάζονται όλοι μαζί και καλύπτοντα βαθμία όλη την Ευρώπη θα καταλήξουν τελικά να είναι πάροχοι υπηρεσιών πανευρωπαϊκοί. Η κυρία Φώστερ τώρα έχει πάρει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση για την κυρία Κρίντ. Όσον αφορά την πρόταση για τα οδικά τέλη, το βασικό ζήτημα είναι να δούμε αν η πρόταση αυτή συνάδει τελικά με την αρχή της επικουρικότητος. Πιστεύετε ότι πραγματικά θα πρέπει να αναλάβουμε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιλύσουμε προβλήματα όπως η συμφόρηση. Προβλήματα τα οποία έχουν σαφώς τοπική και περιφερειακή φύση και πολλές φορές διαφορετικές τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν αναφέρθηκα αυτή τη στιγμή στο ζήτημα της εσωτερήκευσης του εξωτερικού χρέους. Όσον αφορά όντως τη συμφόρηση, και την αντιμετώπιση της, νομίζω πραγματικά ότι όντως μπορούν να υπάρξουν καλύτερες λύσεις σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το τέλος αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Πολλές φορές υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο εμφανίζεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Διαφορετικά θα αντιμετωπιστεί λοιπόν στο Λονδίνο ή στα μεγάλα αστικά κέντρα και διαφορετικά σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου. Για παράδειγμα αυτοκινητόδρομοι που χρησιμοποιούνται από πάρα πολλούς εργαζόμενους σε συγκεκριμένε περιόδους της ημέρας, π.χ. για να πάνε στη δουλειά τους. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση ακόμα πάλι για εσά. Συμφωνείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αναγνώριση στην πρόταση αυτή για το αν μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται σε αστικές περιοχές ή σε περιοχές της υπαίθρου. Πολλές φορές οι άνθρωποι που ζουν στην Ήπεθρο αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους. Μπορούν εν μέρη να επαφίονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στους σιδηροδρόμους, αλλά και πάλι χρειάζονται πάντα και πολύ περισσότερο το αυτοκίνητό τους. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν ε, έχει ε, προνοήσει αρκετά η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτού και τελικά ενδεχομένω να καταλήξουν ιδιαίτερα ζημιωμένοι. Αναφέρομαι σε ανθρώπου όπω οι αγρότε που συμβάλλουν πάρα πολύ στην οικονομία των χωρών του. Όντω, ε, οι δαπάνε είναι αρκετά υψηλέ για τα νοικοκυριά και για τα νοικοκυριά εκείνα που ζουν στην Ήπεθρο. Όχι μόνο η πρόταση αυτή θα είναι επιζήμια και δαπανηρή, αλλά α μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να αποτελούν τμήμα αυτού που ονομάζουμε mobility mix και δεν θα πρέπει να θεωρούνται μια ξεχωριστή κατηγορία η οποία θα, θα ζημιώνεται από την πρόταση αυτή και ουσιαστικά θα φαίνεται σαν να τιμωρείται από την πρόταση αυτή. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να προνοήσουμε και για αυτούς. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια ακόμα ερώτηση, μας λέει ότι θα πρέπει να μην έχουμε διακριτική μεταχείριση για τους αλλοδαπούς οδηγούς οχημάτων και ολοφορείων. Θεωρείτε ότι ε, η πρόταση αυτή είναι απλώς μια ευρωπαϊκή πρόταση προκειμένου να επιληθεί ένα πρόβλημα καθαρά εθνικό, το πρόβλημα της Γερμανίας συγκεκριμένα δηλαδή. Ξέρετε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε δράση πέρυσι κατά της γερμανικής κυβέρνησης όσον αφορά το σύστημα διοδίων που έχει. Απάντηση σε καμία περίπτωση ένα εθνικό σύστημα διοδίων δεν θα πρέπει να εισάγει κριτική μεταχείριση κατά των ξένων χρηστών. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Λεβισκάτορ. Έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, προς την κυρία Κρέτη συμφωνείτε ότι ο αντίκτυπος της έλλειψης διαλειτουργικότητας και για τις επιχειρήσεις και για τους ιδιώτες διαφορετικά διόδια, διέλευση συνόρων κτλ. είναι ουσιαστική, ουσιαστικός. Ναι, είναι ένα ζήτημα, αλλά είναι δύσκολο να συγκρίνουμε ένα σύστημα μόνο για τις μεταφορές με ένα άλλο. Ναι, αλλά είναι σημαντικός ο αντίκτυπος, συμφωνείτε. Επομένως, υπάρχει τρόπος να επιτύχουμε διαλειτουργικότητα χωρίς την νομοθετική πρόταση, ανεξαρτήτως των ε, τροπολογιών που θα ενέχονται. Θα υπήρχε άλλη δυνατότητα και ποια θα ήταν αυτή για να επιτύχουμε τη διαλειτουργικότητα. Να διαθέσουμε το πλαίσιο και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν διακρίσεις. αναλογικά τέλη, αναλογικά σήματα τέλους, οδικά τέλη, διόδια και... Εκτός μικροφώνου ο μιλητής τώρα. Ναι, αυτό σχετίζεται με αυτό που είπατε. Το earmarking είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να το επιβάλλει κανεί στα κράτη-μέλη. Και στο παρόν σύστημα φαίνεται να είναι ανεπαρκές. Εννοείται, όχι μιλώ για την διαλειτουργικότητα, όχι για την χρηματοδότηση. Θα επιτύχουμε τελικώς το, το στόχο μας ή όχι. Αν πετύχουμε μία συστηματοποίηση, όταν υλοποιηθεί θα υπάρχει μια διαλειτουργικότητα για τους πολίτες χωρίς να πιέζουμε υπερβολικά προς την χιλιομετρική επιβάρυνση. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κούλονεν, είχατε ήδη από πριν δικαίωμα από πριν, τώρα σας δίνω τρία λεπτά και μετά θα σας δώσω άλλα τρία αργότερα. Τρία λεπτά κυρία Κούλονεν. Μια ζητώ συγγνώμη αλλά ήμουν μεταξύ άλλων επιτροπών αυτά αντιμετωπίζω καθημερινά. Για τα διαλειτουργικά συστήματα τα συστήματα χιλιομετρικής και άλλης επιβάρυνσης στα διάφορα κράτη θεωρείται ότι υπάρχει μια δυνατότητα τεχνολογικά να βρούμε μια λύση στα σημεία διέλευση των συνόρων π.χ. χωρίς να υποχρεώσουμε τα κρατη να αλλάξουν τα δικά τους συστήματα τελών προς πανευρωπαϊκά συστήματα. Και άλλη μια ερώτηση, η χρησιμοποίηση των εσόδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από, δηλαδή των εσόδων των διοδίων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια 7 ώστε να οικοδομούνται και χώροι ανάπαυσης στο δικοδίκτυο. Ε, ναι, κυρία μου, σε ποιον ε, θέτετε το ερώτημα. Μόλις φτάσατε κατανοώ, αλλά πρέπει να διευκρινίσετε. Φαντάζομαι ότι το πρώτο σας ερώτημα απευθύνεται στον κύριο Μπενεντέτο και τον κύριο Διονέλη, στους φορείς τέλος πάντων. Και το δεύτερο ενδεχομένως στο ERU, δεν ξέρω. Να θεωρήσω αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσει ο κύριος Μπενεντέκτο, εμπαστώση. Μάλιστα, πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι περισσότερο θέμα τεχνολογίας η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Έχουμε τέλη που μπορούν να υπολογίζονται ανάλογα με τα, πόσα, με τα όσα προβλέπει η οδηγία της Ευρωβινιέτας ή χιλιομετρικά. Αλλά πρέπει να είναι σαφές το input και τελικά το άχθος. Η δορυφορική τεχνολογία θα μας επέτρεπε σήμερα να έχουμε συνολική διαλειτουργικότητα των εσόδων. Ο κύριος Διονέλης. To build up... Ε, κοιτάξτε, η τεχνολογία μπορεί να δώσει όλες τις λύσεις. Μπορούμε να έχουμε διαλειτουργικότητα σε όλη την Ευρώπη, αλλά το κόστος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αν το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό, τότε οι, φορεί, οι φορείς της αγοράς δεν θα προσέλθουν. Αν ξεκινήσουμε από διαλειτουργικότητα μεταξύ δύο κρατών, υπάρχει ένα κόστος. Μεταξύ τριών, ακόμα περισσότερο. Και τα λοιπά. Όλο αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό δηλαδή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ για τη δεύτερη ερώτηση για τις υποδομές, τους χώρους ανάπαυσης κτλ. Ίσως ο κύριος Λεμπεντά θα ήταν ο κατάλληλος να σας απαντήσει. Κοιτάξτε, τα έσοδα των διοδίων και των τελών για να χρηματοδοτήσουμε χώρους στάθμευσης ή ανάπαυσης είναι κάτι που εμείς το υποστηρίζουμε απολύτως αυτό. Δηλαδή συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κυρία Κούλωνεν. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε στην κυρία Κούλωνεν για τα επιπλέον τρία λεπτά σας. Νταλουντέ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει κανείς να αμφισβητήσει τον σοσιαλισμό των οδών και να δεχθεί την οικονομία της αγοράς στους δρόμους. Πρέπει ο Ριπένον να πληρώσει, να αναλάβει τις ζημιές, πρέπει να εξωτερικοποιήσουμε το κόστος Ανάλογα με την αρχή αυτή, θέλουμε χιλιομετρικό άχθος ε, για τα φορτηγά, χρειαζόμαστε έντονο τέλος για τον άνθρακα και χρειαζόμαστε ένα μπόνους μάλλον σύστημα αγοράς οχημάτων. Ανάλογα δηλαδή με την περιβαλλοντική επίδοση των οχημάτων. Επομένως η ερώτησή μου είναι, γιατί πρέπει να μείνουμε σε ένα σοβιετικού τύπου σύστημα υψηλή συμφόρησης και ρήπανσης, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ένα σύγχρονο σύστημα της αγοράς που να χρησιμοποιεί λιγότερους δημόσιους πόρους και να δίδει περισσότερα κίνητρα για καθαρή χρήση. Σε ποιον είναι το ερώτημα, λέει ο Πρόεδρος. Σε όσους εκφράζουν αμφιβολίες για ένα σύστημα της αγοράς Προφανώς σε μένα πάει το ερώτημα, λέει η κυρία Κρίντ. Καταρχάς θέλουμε κινητικότητα. Θέλουμε μια κοινωνία που να μπορεί να αναλάβει το κόστος της μετακίνησης. Για την εξωτερήκευση του κόστους, χιλιομετρική ε, επιβάρυνση κτλ. Θέλουμε ισότιμη μεταχείριση γιατί πολλά από αυτά που λέτε για το τέλος για τον άνθρακα ε, το κάνουμε ήδη. Επομένω, έχουμε διαφορετική ερμηνεία ή κατανόηση του τι είναι το επιθυμητό επίπεδο τη φορολόγηση εδώ. Ε, συμφωνώ, λέει ο κ. Λεμπεντά, αν μπορώ να, με αυτά που λέτε, αν μπορώ να προσθέσω, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο τι αποφασίζουμε ότι είναι καθαρό ή όχι. Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, τα ηλεκτρικά, είναι καθαρά εξορισμού. Αλλά πώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. Αν την παράγεται από άνθρακα είναι καθαρή. Επομένως ε, επανέρχεται το ερώτημα. Σας το επιστρέφω δηλαδή. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι η Σουηδική κυβέρνηση είναι στην τελική φάση προετοιμασίας ε, πρότασης για χιλιομετρική επιβάρυνση σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς δείκτες. Έχετε κάποια συμβουλή για εμάς στη Σουηδία για το πώς θα υλοποιήσουμε τη μελλοντική διαλειτουργικότητα. Ναι, λέει ο κ. Διονέλης. Καταρχάς πρέπει να διαρρέσετε δύο, τις δύο αρχές. Ο ρηπαίνων πλεώνει και ο χρήστης πλέον. Αυτό, η πρώτη πρέπει να ε, καλύπτεται. Το ένα τμήμα των εσόδων δηλαδή και του κόστους. Το άλλο, εξωτερικό κόστος, πρέπει να αμφασίζεται σύμφωνα με τη χώρα σας, τι ποσοστό θέλετε να καλύψετε και πού θα χρησιμοποιήσετε τα έσοδα από αυτήν την εσωτερήκευση. Merci Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γιούτο τώρα έχει το λόγο για δυόμιση λεπτά. Κυρία Γιούτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς τον κύριο Τότσε. Όσον αφορά τα διόδια, είπαμε ότι δεν είναι απαραίτητο ότι τα έσοδα από τα διόδια θα πρέπει να επαναπενδύονται στο δικό δίκτυο στι μεταφορέ, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τη χρηματοδότηση σχολείων, νοσοκομείων κτλ. Άρα ουσιαστικά επιβάλλουμε ένα επιπλέον περιβαλλοντικό κόστο χωρί να κάνουμε όμω τίποτα ουσιαστικά για το περιβάλλον, έτσι δεν είναι. Ενώ ο στόχος τελικά της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος θα μπορούσε ουσιαστικά να α, καλυφθεί με το κόστος αυτός, έτσι δεν είναι. Και όσον αφορά τις ανάγκες της αγοράς, μπορούν αυτές να ισχύσουν στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, να καλυφθούν δηλαδή. Κοιτάξτε, όσον αφορά το earmarking, σε έναν βαθμό μπορούμε να πούμε ότι είναι θεωρητική λίγο η ερώτηση, γιατί όσες χώρες έχουν τέτοιο σύστημα δική τιμολόγηση έχουν πάντα χρήματα που επιστρέφουν τελικά στο δικό δίκτυο. Αυτό βλέπουμε τελικά στο Βέλγιο έχουμε οδηγηθεί εκεί πέρα σε μια κάποια αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα μπορεί να γίνει υποχρεωτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι είναι αναγκαίο, ούτε θα ήταν εφικτό. Το έχουμε, κάνει, το έχουμε συστήσει αυτό πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν. Το δεύτερο ερώτημά σα μπορεί να επαναλάβετε, σας παρακαλώ. Ναι. Όσον αφορά το ΜΑΡΚΑΠΑ, αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αυτό το περιθώριο κέρδους δηλαδή, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σας, το συγγνώμη. Όταν λέτε Up, σε τι αναφέρεστε ακριβώς. Ναι, αυτό το επιπλέον κόστος ουσιαστικά πού μπορεί να εφαρμοστεί, πού μπορεί να επιβληθεί. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, πρέπει να επανέλθω στο ερώτημα αυτό αργότερα, αν το επιτρέπετε. Κάτι ακόμα. Έχω λίγο χρόνο ακόμα κύριε Πρόεδρε. 20 δευτερόλεπτα κύριε Αιούτο. Στον κύριο Μπενεντέτο θέλω ουσιαστικά να αποτανθώ, εκτός μικροφώνου. Τα όσα είπατε για τη δορυφορική τεχνολογία. Για ποιο λόγο να μην αρχίσουμε ήδη από τώρα να εφαρμόζουμε τη νέα αυτή τεχνολογία και για ποιο λόγο ουσιαστικά να το αφήσουμε για το μέλλον, έτσι δεν είναι, αν μπορούμε από τώρα. Μα απάντηση, γιατί θα ήταν ακόμα πιο ακριβό να αρχίσουμε ήδη από τώρα να εφαρμόζουμε τη νέα αυτή δορυφορική τεχνολογία. Πάντω, είναι σίγουρο ότι προϊόντος του χρόνου τα αυτοκίνητα θα είναι όλο και πιο στεδεμένα, άρα αργά ή γρήγορα θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη νέα αυτή δορυφορική τεχνολογία όλο και περισσότερο. Κυρία Αγνοτού έχει το λόγο για δυόμιση λεπτά τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ αντίθετα με πολλούς συναδέλφους θεωρώ ότι η βελτίωση όλων των υποδομών και των οδικών υποδομών θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, σεβόμενη παράλληλα βέβαια και την αρχή της επικουρικότητας. Κύριε Ρικέ, εγώ είμαι λιγότερο αισιόδοξη, γιατί βλέπω ότι τελικά το πιο σημαντικό είναι να δούμε ποιος θα πληρώνει και πού θα πηγαίνουν όλα αυτά τα έσοδα. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται εις βάρος του Γάλλου ή του Ευρωπαίου φορολογούμενου και σίγουρα όχι εις βάρος των οδηγών, έτσι δεν είναι. Θα ήθελε επίση ο κύριος Διονέλης να με καθησυχάσει σε κάτι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είπατε ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελεκτρονικών Διοδίων να αναπτυχθεί. Να γνωρίζουμε όμως πού θα εφαρμόζεται και ποιος θα πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένα ποσά σε συγκεκριμένε αρχέ. Νομίζω ότι τίθεται ένα ζήτημα προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ω προ αυτό, τι κάνουμε, τι εχέγγυα μπορείτε να μα δώσετε. Κοιτάξτε, εγώ το αντίθετο είπα. Είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολιτικό όραμα για να φτάσουμε στο στόχο που περιγράψατε, δεδομένης όμως της υφιστάμενης πραγματικότητας, θεωρώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε σταδιακά και βαθμία. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες μικρές περιοχές και περιφέρειες για να δούμε πώς λειτουργεί η λειτουργικότητα επιτόπου, που εντοπίζονται δεχομένως προβλήματα σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα απορρίτου και ιδιωτική ζωή που θέσατε, να δούμε επίση ποια θα είναι οι παράγοντε τη αγορά, και σιγά σιγά να περάσουμε στο πανευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώ όλοι θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πολύ νωρί για να καταλήξουμε στο σύστημα αυτό και ενέχονται και πάρα πολλοί κίνδυνοι. Συμφωνώ, το κατάλαβα αυτό το σταδιακό το οποίο προτείνεται, αλλά το σταδιακό τελικά θα μας βγάλει που στο πανευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι δεν είναι, εκεί δεν θα καταλήξουμε. Εγώ πιστεύω ότι ενέχεται σημαντικός κίνδυνος και σε αυτή την προσέγγιση. Σας ευχαριστούμε κυρία Γνωτού. Ο κύριος Βίμτε Κάμπ τώρα έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα από, μία από τις ωραίες ερωτήσεις είναι πότε θα είναι έτοιμο το σύστημα αυτό στην Ευρώπη. Και αυτό θέλω να θέσω σε ερώτημα και στους πέντε αμελητές. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί και πότε θα λάβει χώρα. Τι εκτιμάτε. Να ξεκινήσω με, το, με τον κύριο Μπενεντέτο. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα εξισορρόπησης του κόστους με τις επενδύσεις και της ετοιμότητας ε, των χρηστών. Δεν μπορώ να κάνω προβλέψη χρονική αυτή τη στιγμή. Προφανώς και εγώ θα πάω στην ε, διαδικασία βήμα προς βήμα να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες των κρατών μελών και πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα αυτά θα είναι λειτουργικά προκειμένου σε όλες τις φάσεις να είναι τα συστήματα και να είναι εύκολα στη χρήση σεβόμενοι τις αρχές. Ε. Βασικός ε, σκοπός είναι να αποφύγουμε την αθέμητη ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων και των κρατών μελών. Όσοι είναι έτοιμοι να καταστούν παροχή ETS ε, και να παρέχουν υπηρεσίες σε όλα τα, όλους τους χώρους διαδίων. Όταν θα υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, η αγορά από μόνη τη θα προχωρήσει. Ω σιδηρεοδρομή, προφανώ ε, υποστηρίζουμε την αρχή τη διαλειτουργικότητα που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό είναι το προφανέ. Και την ε, το να είναι δίκαια τα συστήματα σε όλους τους, σε όλες τις, ε, τους τρόπους μεταφορών. Για μας ως περιβαλλοντική οργάνωση ο σκοπός είναι να κινηθούμε προς μεγαλύτερη ιστορικοποίηση του εξωτερικού κόστους. Και νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ από τα δεκαετία του 90 και κάθε νέο σχέδιο της Ευρωβινιέτας έχει προκαλέσει βελτιώσεις. Προφανώς ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος και ούτε και η παρούσα το παρόν σχέδιο θα είναι τέλειο. Είναι διαδικασία εν εξελίξη, να σας πω πώς τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Η γεωγραφία των μεταφορών. Φανταστείτε να ξεκινήσουμε με την πρώτη περιφέρεια. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία έχουν την πρώτη περιφερειακή τη και παράλληλα θα υπάρχουν και άλλες περιφερειές, η Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία. Εκεί θα υπάρχει άλλη περιφερειακή τη Μετά θα πάμε στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη και έτσι θα έχουμε περιφερειακές, τρεις περιφερειακές ε, Όταν αυτά λειτουργούν, εντάξει, όλα καλά, αλλά το επόμενο βήμα προφανώς θα είναι αυτή η περιφερειακή διαλειτουργικότητες να γίνουν πανευρωπαϊκές. Αυτό θα πάρει χρόνο. Αλλά ξεκινήσουμε πρώτα από το προφητικό επίπεδο. Και ποιο έτος έχετε υπόψη σας. Πότε, πότε. Ποιο έτος. Κι εγώ, ναι, τώρα, δεν λέω, αλλά πότε. Να ακολουθήσουμε τις περιφερειακές διαλειτουργικότητες. Όταν αυτές εμφανιστούν, τότε θα έρθει η ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα. Όχι, θέλω να μου πείτε το έτος συγκεκριμένα, λέει ο κ. Δεν ξέρει, σα λέμε. Το λόγο έχει ο Καπούτο για τρία λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Α αποφύγουμε τι ερωτήσει που έχουν ήδη γίνει από του συναδέλφου. έτσι δεν είναι, όσον αφορά, για παράδειγμα, τη διαλειτουργικότητα. Μία ερώτηση προς τον κύριο Μπενεντέτο. Όσον αφορά το σύστημα αυτό ανάγνωσης των πινακίδων. Προβλέπεται στο νέο αυτό σύστημα ότι θα μπορεί αυτό να γίνεται και με τρόπο αυτόματο, αυτόνομο, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται πιο εύκολα και αυτόματα το όχημα. Η τεχνολογία αυτή αναγνώρισης των πινακίδων θεωρείται ένα μέτρο συμπληρωματικό σε σχέση με άλλες τεχνολογίες και ότι θα πρέπει να υπάρχει σε σχέση με άλλες ε, υπηρεσίες όπως για παράδειγμα τηλεδιόδια και καταβολή άλλων οδικών τελών. Όπου έχει χρησιμοποιηθεί αυτόνομα και ξεχωριστά δεν έχει δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πιστεύετε εσείς ότι στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος ε, ηλεκτρονικών διοδίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό αναγνώρισης ε, των πινακιδών και να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα και ξεχωριστά ή θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με τα άλλα συστήματα. Κοιτάξτε, το μέσο αυτό στο οποίο αναφερθήκατε αποτελεί ένα καταπληκτικό συμπληρωματικό σύστημα και ένα σύστημα backup αναδίπλωσης δήλω. Δηλαδή, αν ε, χρειάζεται να εντοπιστεί ένα συγκεκριμένο όχημα. Αυτή τη στιγμή το σύστημα ανάγνωσης ε, των πινακίδων δεν έχει δώσει ακόμα έμπιστα αποτελέσματα. Ενώ αντίθετα με τα άλλα συστήματα έχουμε πολύ πιο υψηλά ποσοστά όσον αφορά τα αποτελέσματα. Ξέρετε ότι δεν είναι πάρα πολλές φορές εύκολο οι μικρές πινακίδες, τα μικρά οχήματα να αναγνωστούν. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να καταβάλουμε περισσότερες δαπάνες για ένα σύστημα το οποίο τελικά δεν θα είναι αρκετά αποτελεσματικό. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ότι ενδείκνεται μάλλον να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό σε συνάρτηση με άλλες τεχνολογίες, έτσι δεν είναι ακριβώς, ναι. Μια άλλη ερώτηση τώρα προς τον κύριο Τόντ. Κάτι το οποίο κάλυψαν εν μέρη και άλλοι συνάδελφοι όσον αφορά την τιμολόγηση, την κοστολόγηση, τον καθορισμό της κοστολόγησης δηλαδή σε σχέση με τις ε, επιπτώσεις τις περιβαλλοντικές. Να ασχοληθώ με μια συγκεκριμένη διάσταση του ζητήματος, το ζήτημα της διαφάνειας και της κοινοποίηση προς τον ε, καταναλωτή, προς τον χρήστη. Θα ήθελα με άλλα λόγια να καταλάβω αν συμφωνείτε κι εσείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση και μια καλύτερη επικοινωνία προς τον τελικό χρήστη Πώς καθορίζονται δηλαδή τα ποσά τα οποία καλείται να καταβάλει στα πλαίσια των οδικών τελών. Για ποιο λόγο πρέπει να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Πιστεύετε ότι η καλύτερη αυτή ενημέρωση θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο τελικά χρησιμοποιούμε τα μέσα μεταφοράς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και για παράδειγμα, η διαφοροποίηση Euroclass που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ακριβώ αυτό το μήνυμα και πραγματικά έχει βοηθήσει να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο οχήματα τη τάξη Euro 6. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και για το σύστημα αυτό των τηλεδιοδίων, το πανευρωπαϊκό, να μπορούμε να έχουμε ακριβώς την ίδια ταξινόμηση. Για 1,5 λεπτό τώρα το λόγο έχω εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Προς τον κύριο Λόκμαν ως προς το earmarking. Αν το earmarking ε, μπορεί τελικά να χρησιμοποιείται και για τις οδικές μεταφορές αλλά και για άλλους τρόπους μεταφοράς, τους σιδηροδρόμους για παράδειγμα. Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε ποιο ποσοστό θεωρείτε ότι θα ήταν εύλογο να χρησιμοποιηθεί. Στο earmarking αναφέρομαι. Κοιτάξτε, όπως σας είπα ήδη, το earmarking νομίζω ότι συνδέεται ουσιαστικά με την επιβολή των οδικών τελών υπέρ της αναβάθμισης υποδομής. Όσον αφορά τα markups τώρα, οι προσαυξήσεις αυτές, τα επιπλέον τέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη καθαρών μορφών μεταφοράς. Και όσον αφορά την αρχή ο πληρώνει, αυτή είναι μια δαπάνη που θα πρέπει ουσιαστικά να αποτελέσει αντικείμενο εσωτερήκευσης, εξωτερικό κόστος που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εσωτερήκευσης. Ναι, αλλά όσον αφορά το marketing. πιστεύετε ότι μπορεί να αφορά παράλληλα πολλούς διαφορετικούς τρόπους μεταφορών, όχι μόνο τις οδικές δηλαδή μεταφορές. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει σε κρατικό επίπεδο να το μελετήσουμε. Άρα δεν μπορώ να μου απαντήσετε τώρα, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Ο κύριος Βίμπαντεκάμ πάλι θέλει το λόγο. Δεν θέλετε το λόγο, σα αντιστοιχούσαν τρία λεπτά από το ΕΛΚ. Δεν τα θέλετε. Πολύ ωραία. Η κυρία Κίλονεν τότε πάλι. Έχετε κι εσείς τρία λεπτά. Κυρία Κίλονεν, παρακαλώ. Έχετε τρία επιπλέον λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Από την κυρία του πάνελ θα ήθελα να καταλάβω ποια θα ήταν η λύση σας να ξεκινήσουμε επί να ξεκινήσουμε από το μηδέν για τα οδικά τέλη. Και πάλι θα έπρεπε να προσαρμοστούμε σε εθνικές ανάγκες και συνθήκες. Επικορικότητα σε εθνικό επίπεδο λοιπόν. Και κάτι από αυτά που βρίσκουμε δύσκολα ως ενώσεις μεταφορέων κάθε χι χρόνια άλλη μια τάξη οχήματο θεωρείται καθαρό ή καλύτερο ή πιο καθαρό, οδηγούμαστε προς μια κατεύθυνση και μετά αποδεικνύει ότι δεν ήταν έτσι. Είτε αυτό αφορά στους σιδηροδρόμους, είτε στα ηλεκτρικά οχήματα, είτε οτιδήποτε. Η, η τεχνολογία, η επιστήμη αλλάζει τα ευρήματά της. Και αυτό που θεωρούσαμε καθαρό μέχρι πριν μπορεί να μην είναι καθαρό αύριο. Επομένως εμείς το βλέπουμε από, υπό την οπτική του χρήστη. Δεν υπάρχουν ούτε διάβολοι ούτε άγγελοι. Ε, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που σας παρέχουν διαφορετικές λύσεις. Αν έχετε εκπτώσεις για τα ηλεκτρικά, ηλεκτρικά οχήματα στους αυτοκινητοδρόμους, αυτό δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό από την έννοια του κόστου ωφέλους, γιατί δεν, είναι καθόλου δεν κινούνται επαρκώς ε, γρήγορα. Επομένως το τι αποδέχεται κανείς, το ποιο είναι αποδεκτό, είναι κατά πόσον οι κυβερνήσει επιτυχάνουν τους στόχου που θέτουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αυτό με καλύπτει απολύτω, ως απάντηση, λέει η κυρία Κούλονεν. Τέλεια, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκραπίνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα και θα ήθελα και σύντομες ε, απαντήσεις παρακαλώ. Κάποιοι θέλουν τα σήματα τέλους, άλλοι δεν τα θέλουν, κάποιοι θέλουν επικορικότητα, άλλοι δεν θέλουν. Αντιφατικά όλα αυτά. Η κυρία Κρίντ, για τη φορολόγηση, ποια είναι η συγκεκριμένη σας πρόταση για να είναι δίκαιη αυτή η επιβάρυνση. Τι προτείνετε ακριβώς, ώστε τα έσοδα να επανέρχονται στις υποδομές. Με συγκεκριμένη πρόταση. Κύριε Τόντ, είπατε ότι δεν θα ήταν καθόλου ακριβό να χρησιμοποιεί κανείς ηλεκτρονικά οχήμα, ηλεκτρικά οχήματα. Έχετε μελέτη αντικτύπου. Γιατί σε πολλές ε, ζώνες ε, δεν υφίστανται καθόλου και στην Ήπεθρο είναι πολύ λίγο πρακτικό. Πώς θα το επιτυγχάνατε. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει η κυρία Κρίντ. πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ισότιμα. Εγώ δεν θα ήθελα να δαιμονοποιήσουμε τη βινιέτα ότι είναι η πηγή όλων των κακών. Πρέπει όλα να συνδέονται στη χρήση με δεδομένα αποδείξεις του τι είναι η καθαρή χρήση και μην είστε απόλυτα βέβαιοι τι θα είναι το καθαρό αύριο όπως έλεγα. Επίσης, να είστε σίγουροι ότι οποιοδήποτε μέτρο θα είναι κατάλληλο για την εθνική αγορά για τα ηλεκτρονικά οχήματα, λέει ο, ο, αν έχετε ηλεκτρικό όχημα που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια αντί για ντίζελ ή βενζίνη, είναι πολύ πιο φθηνό στη χρήση του. Αν έχουμε όλα και περισσότερα στο μέλλον, αυτό εννοούσα. Είχα... Ε, εννοούσα κάτι τελείως διαφορετικό. για την ε, επιστροφή των επενδύσεων. Στις επενδύσεις αν είχε αναφερθεί ο κύριος Τόντς. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι κάθε κράτος μέλος θέτει διαφορετικές προτεραιότητες. Αν έχει κανείς έσοδα ένα δισεκατομμύριο από τα διόδια, μπορεί κανείς με αυτό να μειώσει το εργατικό του κόστος αν έχει πολύ υψηλό. Τι να σας πω. Ή μπορεί να επενδύσει στο δικό δίκτυο, αλλά είναι μια επιλογή των κρατών μελών. Λοιπόν, ε, έτσι είναι τα πράγματα. Ίσως ε, εκνευριστικό αλλά αληθές η ερώτηση ήταν ευρεία. Λοιπόν, δύο λεπτά για τον κύριο Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε και μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ε. αυτά που είπε η κυρία Γκρίτα και μου δημιουργήθηκε μία ερώτηση. Τι σημαίνει το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει τελικά να επιβαρύνουμε επιπλέον τους χρήστες. Δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τι γίνεται με τα τέλη, τα οποία είναι και πολύ υψηλά. Σωστά κατάλαβα αυτό που είπατε. Ναι, αυτό ε, εννοούσα. Αν και δεν είπα και δεν εννοούσα τις ε, εταιρείε. Εννοούσα ότι αποτελεί αυτό μεγάλο φορτίο για τους πολίτες. Κόστος του χιλιάνα χιλιόμετρο θα ήταν 10,8 cents ε, λεπτά του ευρώ κατά τη διαστολή με τα σημερινά συστήματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Λιμπεράτσκι. Αυτό σημαίνει ότι το πακέτο αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Μια ερώτηση προς τον κ. Πεντέτο. Αυτό το πακέτο μπορεί να είναι πραγματικά ενδιαφέρον, για παράδειγμα, είναι σε κάποιες ορισμένες χρονικές στιγμές τριπλάσια η επιβάρυνση για την ε, κυκλοφορία στους δρόμους των Βρυξελών, για παράδειγμα. Και αυτό προφανώς θα εκκρατηθεί το σύστημα, προφανώς. Ε, όντως, ισχύουν διαφορετικά συστήματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και εμεί ω φορεί παροχή υπηρεσιών πρέπει να είμαστε θέσει να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κατάσταση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία τρίτη ε, ερώτηση, κύριε Μπενεντέτο. Είπατε ότι κατά βάση είσαστε αυτοί που εισπράτεται. οι πελάτες θέλουν ουσιαστικά να πληρώσουν. Αυτό είπατε. Ε, Κοιτάξτε, είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Εμείς ε, εισπράττουμε ουσιαστικά τα χρήματα από τους πελάτες εκείνες που οφείλουν ουσιαστικά ε, ακόμα χρήματα. Υπάρχει και η μέθοδος της πίστοσης αλλά από την άλλη προσπαθούμε να βρούμε και κάποιες ε, διευκολύνσεις. Εμείς πάντως εισπράττουμε τα χρήματα αυτά και με τις συμφωνίες που έχουμε έπειτα με τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις υποδομές των διοδίων φροντίζουμε να διαθέσουμε τα χρήματα αυτά από τους χρήστες προς ε, τους φορείς των υποδομών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τώρα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τρία λεπτά τον κύριο Λιεζουά από την DG Move ο οποίος καλείται μέσα σε τρία λεπτά όμως να μας πει ποια είναι η δικιά του άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Μια γενική παρατήρηση, ποιες είναι οι εντυπώσεις μου, θετικές θα έλεγα. Όσον αφορά τις αντιδράσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί και τις παρεμβάσεις που γίνανε για την οδική τιμολόγηση, Υπάρχουν πολλοί που είπαν ότι η οδηγία για την Ευρωβινιέτα μπορεί πραγματικά να δώσει πολύ σημαντικά κίνητρα και να μειώσει τελικά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό μέσο αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και όσον αφορά την διαλειτουργικότητα των διοδίων και την ανάπτυξη μια ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων, ακούσαμε τι ανάγκε του κλάδου ότι θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνε πιστοποίησης των παρόχων υπηρεσιών, καλύτερη τυποποίηση, καλύτερη ξεκάθαρη κανόνες για την τιμολόγηση. Τώρα, η ε, σταδιακή κατάργηση της Ευρωβινιέτας. Αυτό προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρότειναν και πολλοί σήμερα, όπως ε, η TNE και η ε, CER. Στην πρώτη συζήτηση που κάναμε τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη είχαν κάποιες επιφυλάξεις Θέλω να μπορούν να έχουν ε, την εναλλακτική ανάμεσα σε διόδια και βινιέτα, ακόμα και τα κράτη εκείνα τα οποία έχουν μόνο διόδια αυτή τη στιγμή. Καλείται λοιπόν τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει περισσότερο τη βασική αρχή αυτή των διοδίων στις συζητήσεις που θα γίνουν. Όσον αφορά τα λεωφορεία και τα πούλμαν, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, κυρίως από την IRU, και νομίζω ότι ε, ο εισηγητής ε, για την οδηγία της Ευρωβινιέτας είπε ότι κάτι πολύ σημαντικό, τα πούλμαν χρησιμοποιούν την οδική υποδομή, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξαιρούνται από τα διόδια. Χρησιμοποιούν και φθύρουν... και τα πούλμαν το οδικό δίκτυο όπως και όλα τα υπόλοιπα οχήματα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συμβάλλουν και αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει να προωθήσουμε τα λεωφορεία όταν αυτά αποτελούν μέρος των δημοσίων ε, μεταφορών και στα τέλη Νοεμβρίου θα δείτε ότι θα υποβληθεί μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ανοίξει η αγορά για τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Θα δοθούν νέες ευκαιρίες για τον κλάδο αυτό. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα εξαιρούνται από την καταβολή διοδίων. Τώρα, όσον αφορά την κατανομή των εσόδων που προκύπτουν από την οδική τιμολόγηση, το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, όπω καταλαβαίνετε, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα επιμέρου κράτη-μέλη. Θα έλεγα ότι καταρχά θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι οι χρήστε καταβάλουν συγκεκριμένα τέλη τα οποία θα πρέπει έπειτα να χρησιμοποιούνται σωστά από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε πώς τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο σύστημα μεταφορών Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που δεν δέχονται την κατάτμιση την οποία εμείς προτείνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αν μη τι άλλο, ένα κάποιο επίπεδο διαφάνειας μέσω εκθέσεων που θα μπορούσαν να υποβάλουν τα κράτη-μέλη. Διαφάνεια προς την κατανομή τελικά των πόρων που προέρχονται από την οδική ατιμολόγηση. Και για το σημείο αυτό όμως θα θέλαμε να είχαμε μια υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά είχα να σας πω, ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ για τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές ε, παρεμβάσεις που κάνανε. Σας ευχαριστούμε κύριε Λεζουάν, ευχαριστήσω και εγώ τους συμμετέχοντε στο πάνελ και για τη συμμετοχή τους και για το ότι απάντησαν σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Πρόκειται για την πρώτη συζήτηση που κάνουμε για το ζήτημα αυτό και φαντάζομαι ότι ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές θα καταφέρουν να αντλήσουν πολλά σημαντικά διδάγματα. Και τώρα ξέρετε ότι διανύουμε την εβδομάδα σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Ξέρετε ότι πολλές εκδηλώσεις έχουν ήδη προβλεφθεί στη διάρκεια της εβδομάδας αυτής. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι θα πρέπει με τον έναν άλλο τρόπο όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να συμμετάσχουν στην Αφρικανική Εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ πολύ κάντε ησυχία καθώς αποχωρείτε από την αίθουσα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό προκειμένου να μιλήσουμε για την αερομεταφορές στην Αφρική, ένας κλάδος ο οποίος παρουσιάζει πολύ έντονη ανάπτυξη, μολονότι γνώρισε αρκετά προβλήματα. Προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματά μας λοιπόν έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την DG Move, καθώς επίσης και τον εκπρόσωπο της ΕΑΖΑ, οι οποίοι μόλις φτάσανε. Σας παρακαλώ πολύ αποχωρήστε από την αίθουσα χωρίς να κάνετε θόρυβο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τη Μαριάννα εδώ πέρα για θέματα αεροπορία. Όλα πάνε καλά. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπομπέιν για την ε, πολιτική αεροπορία, εμπορική αεροπορία στην Αφρική. Έχετε το λόγο εξ της DG Move της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Μπορώ να πω ακόμα καλημέρα σε όλους. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα ότι στο πλαίσιο της ε, εβδομάδας αφιερωμένη στην Αφρική εδώ στο Κοινοβούλιο, επιλέξαμε να διοργανώσουμε ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της ε, αφρικανικής ε, αεροπλογίας. Μιας και είμαι στον κλάδο, αυτό προφανώς με χαροποιεί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το θέμα της ασφάλειας ότι αφορά ε, την αεροπλογία στην Αφρική γιατί προφανώς η πιο σημαντική υποδομή που υφίσταται στην ε, αεροπορία δεν είναι τα τέρμιναλς και οι αεροδράδρομοι και η τεχνολογία εχμής. Το πιο σημαντική υποδομή είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια σε όλες τις πτυχές. Ε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να πάρω το λόγο για να μιλήσω για το σκέλος της Αφρικής. μικρή εισαγωγική παρουσίαση μαζί με τους συναδέλφους από την ΕΑΖΑ που επίσης δραστηριοποιούνται έντονα στην Αφρική και έχουμε την τιμή να ηγούμαστε της ε, Σχετικής Επιτροπής για την Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας πω ότι χθες ε, στην Ιγυρία παρευρεθήκαμε και σε ένα συνέδριο του ΙΚΑΟ για την ασφάλεια και αυτό καταδεικνύει πω ο κόσμος δίνει σημασία ιδιαίτερη στην Αφρική. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω τους τρει βασικούς πυλώνε, όπως αποκαλούνται, των δράσεών μα και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να παρακολουθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο την ασφάλεια και ιδιαίτερα στην Αφρική. Έχετε αφενός κάτι καινούριο τα τελευταία χρόνια το σύστημα έγκρισης των TCO των, των παρόχων τρίτων, χώρας, τρίτων χωρών. Δεύτερος πυλώνας ε, το σύστημα Σάλφα Ένα σύστημα ε, τυποποιημένων δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη την Ευρώπη. Το πλεονέκτημα λοιπόν είναι το εξής όταν γίνεται έλεγχος ενός αεροσκάφου στην Πρατισλάβα, γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται ο έλεγχος και στο Ελσίνκι και στην Βαρκελόνη, είτε πρόκειται για ένα αεροπλάνο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. Είναι ίδιος απόλυτα ο τρόπος ελέγχου και προφανώς από ό,τι βλέπετε είναι τεράστιος όγκος πληροφοριών που συλλέγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς ε, τα πάνε οι πάροχοι και τι επιδόσεις συμφωνούν ως Ευρωπαίοι δεν θα πρέπει να καθόμεθα βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε περήφανοι. Γιατί η Ευρώπη πραγματικά έχει τα πιο υψηλά πρότυπα σε όλο τον κόσμο και το σύστημα δουλεύει, είναι πολύ αποβατικό και πολλές χώρες πλησιάζουν και προσεγγίζουν την Ευρώπη για να μπορέσουν και αυτές να χρησιμοποιήσουν το σύστημα το οποίο και είναι δυνατόν γιατί προβλέπεται χώρες που έχουν αναπτύξει τέτοια συστήματα Μπορούν να έρθουν λοιπόν σε επαφή με την Ευρώπη για να χρησιμοποιήσουν και για του δικού του σκοπούς το σύστημα αυτό και γι' αυτό λοιπόν εξασφαλίζουμε σε όλο τον κόσμο να μπορούμε να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει για την αεροπορική ασφάλεια. Δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Αφρική ακόμα που να είναι τμήμα τη οικογένεια ΑΦΑ, αλλά είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί πάρα πολύ την ΕΑΖΑ και το επιδιώκει. Τρίτο στοιχείο τρίτος πυλώνας της εργαλειοθήκης μας σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ασφάλεια. Όπως γνωρίζετε, ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Ασφάλειας, blacklist, μαύρη λίστα. Αλλά προσπαθήσαμε να τον διατυπώσουμε με πιο ε, αισιόδοξο τρόπο. Κατάλογος λίστα αεροπορικής ασφάλειας και πάντα είμαστε περήφανοι να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας και να υποστηρίζετε και να ενισχύετε και εσείς τις εργασίες μας από την Επιτροπή σας. Πρόκειται για τρία εργαλεία τα οποία θεωρούμε ότι μπαίνουν στην ίδια εργαλειοθήκη και ένα από τα καθήκοντα. Ε, μία από τις προκλήσεις αυτές είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα τρία εργαλεία, αυτά τα τρία μέσα λειτουργούν απόλυτα μεταξύ τους, ε, συνεργάζονται ομαλά και απρόσκοπτα μεταξύ τους. Εν συντομία τώρα, για την Αφρική, τώρα σε ό,τι αφορά τον κατάλογο αεροπορικής ασφάλειας, η Αφρική εξακολουθεί να εμφανίζονται πιο συχνά στον κατάλογο αυτό από ότι άλλες περιοχές. Αυτό τι σημαίνει και ιδιαίτερως πριν από κάποια χρόνια η αεροπορική ασφάλεια στην Αφρική προφανώς αποτελούσε πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω λοιπόν τι δράσεις λάβαμε μαζί με τους Αφρικανούς εταίρους μας, προκειμένου σταδιακά να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν έχουμε ακόμα πετύχει τον απότερο στόχο μας, αυτό είναι σαφές, γιατί εξακολουθούν να εμφανίζονται υπερβολικά σε αυτή τη λίστα. Αλλά θα δείτε ότι τα πράγματα έχουν σταδιακά αλλάξει, ιδιαίτερα σε χώρες και πάντα επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία, ιστορία όπου οι αρχές ε, αεροπορίας μπορούν να κάνουν ελεύθερες τη δουλειά τους, γιατί η αρχή ε, αεροπορίας ε, θα πρέπει να έχει ανεξαρτησία, θα πρέπει να έχει μέσα και η ανεξαρτησία στην Αφρική δεν είναι πάντα κάτι το αυτονόητο. Και επίση τα μέσα που έχουν στη διάθεσή του οι αρχέ αυτές, οι αρχέ αυτέ εποπτεία, θα πρέπει να είναι επαρκή. Γιατί σε πολλέ περιπτώσει οι αεροπορικέ εταιρείε είναι πολύ πιο πλούσιε από τι ε, υπηρεσίε επιτηρήσει. Αλλά προφανώ οι υπηρεσίε οι δημόσιε είναι αυτέ που θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης. Στην Ιγυρία, για παράδειγμα, αναγκαστήκαμε να βάλουμε έναν, ε, μια ε, αεροπορική εταιρεία στο κατάλογο, στη μαύρη λίστα. Ε, και τότε ξύπνησαν λίγο οι αρχές, οι δημόσιες, οι οποίες κάπως είχαν εφιστεχαστεί και δραστηριοποιήθηκαν. Βλέπετε λοιπόν ότι η Αφρική Εμφανίζεται πολύ συχνά και το σημείο 3 είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουμε τη Ζιμπάμπουε, την Air Zimbabwe και μια αεροπορική εταιρεία της Νιγηρίας μπήκαν στον κατάλογο γιατί η ΙΑΖΑ απέρριψε για λόγους ασφάλειας την έγκριση τη της CEO. Αν λοιπόν μία αεροπορική εταιρεία ζητά έγκριση TCO με την ΕΑΖΑ και η ΕΑΖΑ απορρίπτει για λόγους ασφάλειας, όχι για διοικητικού λόγους, αλλά για λόγους ασφάλειας, αρνηθεί να χορηγήσει τέτοια έγκριση, προσκαλείται αυτόματα στην Επιτροπή αεροπορική Ασφάλειας και κανονικά ο... η εταιρεία αυτή μπαίνει στην λίστα. Αυτό και έγινε με τους δύο αυτούς παροχού. Αυτό που συνέβη είναι το εξή. Αυτό συνήθω αποτελεί το καμπανάκι του κινδύνου για να ξεπνήσουν οι δημόσιε αρχέ τη εκατότητα χώρα ότι κάτι θα πρέπει να κάνουν για να βελτιώσουν την ασφάλεια. Ιδάλλως θα καταλήξουν όλοι ουσιαστικά οι αερομεταφορεί στο κατάλογο αυτό. Εδώ βλέπετε ένα μικρό διάγραμμα, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά καταδεικνύει ιδιαίτερα προ τα αριστερά ότι τα αριθμητικά στοιχεία σταδιακά μειώνονται αργά αλλά σταθερά. Η Αφρική ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και βλέπετε ότι και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αεροπορικών εταιριών και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των χωρών, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια σταδιακά και βαθμία η κατάσταση βελτιώνεται. Δεν ε, δρούμε ελαφριά την καρδιά. Ξέρετε ότι μόνο αν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι έχει πραγματικά με βιώσιμο και μόνιμο τρόπο βελτιωθεί η κατάσταση, μόνο το διβγάζουμε από τον κατάλογο της ασφαλείας. Αυτό μέχρι το 2014-2015 δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν ήμασταν σε θέση, ειλικρινά. Αλλά τώρα συμβαίνει πραγματικά αυτό και το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και συστήνουμε επίσης και στις εταιρείε τι να κάνουν και στις αρχές. Αν λοιπόν ε, αντιδράσουν ακαριέα και αποφασιστικά, εμείς από πλευράς μας είμαστε έτοιμοι να τους βγάλουμε από τον κατάλογο. Αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει το γράφημα αυτό, το διάγραμμα αυτό. Και τώρα βλέπετε μια σύντομη επισκόπηση του τι συνέβη και πώς διαμορφώθηκε αυτή η θετική τάση που καταδεικνύει ότι στο σύνολό της η αφρικανική ασφάλεια αεροπορίας δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι, αλλά σαφέστατα ε, βρίσκεται σε μια θετική ενωδική τάση. Εξέρονται κάποιε ε, χώρες οι οποίες κατρακυλούν. Ε, η Ζιμπάμπουε, για παράδειγμα, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Άλλε χώρε όμω η Μαυριτανία, η Σουαζιλάνδη, η Ζάμπια, ήταν σε θέση να εργαστούν σωστά και καταφέραμε να τις βγάλουμε από την λίστα. Και, όπως σας είπα, σε διάφορες περιπτώσεις χρησιμοποιήσαμε την ε, λίστα και να εντοπίσουμε τις χώρες οι οποίες ναι μεν ακόμα δεν έχουν μπει στη λίστα, αλλά κατρακυλούν και τους βάζουμε κάπως σε το δίλημα ότι είτε θα αναλάβετε δράση και θα επενδύσετε ή ξέρετε πού θα καταλήξετε αυτή η σκιά όπως τη λέμε της λίστας αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αν θέλετε εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Δεν θα επαναλάβω όσα ήδη είπα για τις, ε, τα συστήματα των τρίτων χωρών, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΑΖΑ. Αυτό που διαπιστώνουμε στο σημείο αυτό είναι ότι η ΕΑΖΑ στο σύστημα αυτό το οποίο έχει καταστεί λειτουργικό πλήρως μόνο εδώ και δύο χρόνια έχει 19 αφρικανικές εταιρείες με εταιρείε που έχουν λάβει έγκριση DCO από την ΕΑΖΑ. 63 είναι οι εταιρείε που μπορούν να πετάξουν προς την Ευρώπη, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια από τα χρειάζεται τα αξιολόγηση ασφάλειας από την ΕΑΖΑ πρωτού ξεκινήσουν οι πτήσεις προς και από την Ευρώπη. Αυτό δεν ίσχυε, γιατί ήταν εθνικά τα προγράμματα στο παρελθόν. Άρα όποιοι υποβάλλουν τέτοια αίτηση θα πρέπει να πληρούν πρότυπα ασφαλεία τα οποία να τα έχει εγκρίνει η ΕΑΖΑ. Πρωτού ξεκινήσουν οι πτήσει προ την Ευρώπη. Προφανώ αυτό αποτελεί χρήσιμο, ωφέλιμο και ενδιαφέρον στοιχείο. Στη συνέχεια, ένα αριθμό εταιριών ε, ε, κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα επιθεώρησης του αεροσκάφους. Το ονομάζουμε σύστημα ΣΑΦΑ και δεν θέλουμε να το αλλάξουμε, μας αρέσει αυτό το όνομα. Αυτό που θέλουμε να ξέρουμε είναι ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε κατά πόσον ε, πληρούνται και εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα, γιατί ξέρουμε ότι σε κάποιους τομείς τα ευρωπαϊκά πρότυπα υπερβαίνουν τα διεθνή και πολύ σωστά κάνουν, αλλά η εταιρείε τρίτων χωρών ουσιαστικά εμ, πρέπει να πληρούν τα διεθνή πρότυπα τα οποία τα προδιαγράφει ο ΙΚΑΟ. Και οποιαδήποτε κράτος υπό τη συνθήκη του Σικάγο έχει το δικαίωμα να διεξαγάγει τέτοιες επιθερήσεις. Όπως σας είπα, οι τρίτες χώρες έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν στο σύστημα. Η Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, ο Καναδάς, η Αυστραλία έχουν ήδη προσχωρήσει και μερικές άλλες χώρες. Και το πιο ενδιαφέρον σύστημα είναι ότι στο παρελθόν γνωρίζαμε ότι αυτό συνέβαινε και ουσιαστικά κάποιες αεροπορικές εταιρείες έκαναν, <coughs> έστελναν πιο καλά πληρώματα, τα πιο καλά αεροσκάφη στην Ευρώπη. Γιατί, γιατί ήξεραν ότι στην Ευρώπη θα αντιμετώπιζαν τους πιο αυστηρούς ελέγχους. Αυτό τι σήμαινε ότι τα χειρότερα πληρώματα και τα χειρότερα αεροσκάφη κατέληγαν αλλού τώρα αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο φυσικά να υλοποιηθεί γιατί και αλλού θα έχουν τα πρότυπα σάφα για παράδειγμα. Δεν θα είμαι διπλωματικός. Ε. Ε, πλέον τα χάλια αεροπλάνα δεν τα στέλνουμε στη Μέση και τα καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, ξέρουν ότι αν ε, και στον Περσικό κόλπο και στην Ασία και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική θα τους εντοπίσει το σύστημα και ότι κάθε εταίρος του συστήματος θα λάβει τις πληροφορίες από τις υπόλοιπε επιθεωρήσεις που έχουν διεξαχθεί για κάθε εταιρεία. Και πάλι πρέπει να σας πω ότι στην Ευρώπη δεν συνειδητοποιούμε ότι συστήνουμε συστήματα στην Ευρώπη τα οποία τα ζηλεύει ο υπόλοιπο κόσμο. Και με την υποστήριξή σα στο παρελθόν καταφέραμε να αναπτύξουμε όλα αυτά τα συστήματα. Δεν θα υπησέλθω σε λεπτομέρειε την ε, διαφάνεια αυτή. Αν δείτε στο δεξί τμήμα της διαφάνειας όπου έχουμε την Αφρική, είναι ακόμα η περιφέρεια ε, με τους ε, χειρότερους λόγους ΣΑΦΑ αλλά θα βλέπετε ότι κατέρχονται. Δηλαδή πριν από λίγα χρόνια ήταν πολύ πιο ψηλό το γράφημα. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει σαφής βελτίωση. Ε, το σύστημα επιθεωρήσεων των διαδρόμων απογείωσης και προσγείωσης μας παρέχει πολύτιμα δεδομένα και για τον κατάλογο TCO. Ο κατάλογος αυτός των ε, ξένων αερομεταφορέων λειτουργεί πάρα πολύ καλά και στην Αφρική έχουμε αερομεταφορείς που τα κατάφεραν, που έκαναν, κατέβαλαν προσπάθεια να μπουν στον κατάλογο, να λάβουν δηλαδή την πιστοποίηση και αν ένα μεταφορέας ή μια χώρα θέλει να επιτύχει αυτό το καθεστώς πρέπει να βελτιώσει το επίπεδο ασφαλείας της. Αυτό είναι θετικό για όλους. Επίση, οι αρχές δεν επιθυμούν να αποτύχουν στη δοκιμή TCO οι αερομεταφορεί του και επομένως ε, ε, ασκούν και αυτή πίεση Θα δώσω τώρα το λόγο στον Λουκ Τίτγκατ που είναι διευθυντής ε, για μια σειρά, υπεύθυνος για μια σειρά από πράγματα στρατηγικής σημασία και θα επανέλθω με μια τελευταία διαφάνεια αν μου επιτρέπετε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θα έχετε λάβει όλοι για τα, της λειτουργίας προκειμένου να έχουμε συνθήκες ασφαλείας. Η παρουσία του Πίτερ εστιάστηκε στους ε, μεταφορείς. Εγώ τώρα θα εστιαστώ περισσότερο στο ρυθμιστικό επίπεδο, δηλαδή την αρμοδιότητα των ε, κρατών προκειμένου να έχουμε επαρκή έλεγχο του κλάδου. Ε, χρειάζονται λοιπόν και οι δύο εικόνες για να έχουμε πλήρη εικόνα. Και οι δυνατότητες και συνθήκες ασφαλείας των αερομεταφορέων, αλλά και ότι θα έχουμε δυνατότητα και σε επίπεδο κράτους που φιλοξενούν, κράτη δηλαδή, που φιλοξενούν αερομεταφορείς στις εγκαταστάσεις τους και που ταξιδεύουν από και προς αυτά τα κράτη. Εδώ έχουμε ένα επίπεδο εφαρμογής ε, διεθνών προτύπων ασφαλείας, από κόκκινο που δεν είναι καθόλου καλό μέχρι πράσινο που είναι πολύ καλό. Άρα βλέπετε μια μεγάλη ποικιλομορφία δυνατοτήτων των εθνικών αρχών, μεγάλες αποκλήσεις, Βλέποντας αυτή την εικόνα επίσης αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι εύκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει διότι δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση. Η πραγματικότητα έχει σημαντικές διαφορές. Οι διάφορες χώρες δεν έχουν την την ίδια πρόοδο υλοποίηση διεθνών προτύπων και επομένω δεν υπάρχει ταχεία λύση σε όλα αυτά. Και βέβαια θα ήταν μια συνταγή για καταστροφή στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης ε, της Αφρικής, ε, όπου οι αερομεταφορές είναι σημαντικές έχουμε ένα στοιχείο αυτό της ασφαλείας που θα μπορούσε να το δει κάποια από τις χώρες αυτές, αν αυτό εννοεί ο μιλητής, ως εμπόδιο για την ανάπτυξή της. Επομένως, σε διεθνές επίπεδο πρέπει να δούμε πώς θα προτεραιοποιούμε τις όποιες δράσεις μας. Okay, thank you. So, You Είδατε προηγουμένως μία παρουσίαση και τώρα βλέπετε μία άλλη. Πώς δηλαδή οργανώνουμε τον ΕΑΣΑ ώστε να παράσχει βοήθεια στις εθνικές αρχές. Τα χρώματα εδώ αποτυπώνουν διαφορετικά έργα. Σε γαλάζιο χρησιμοποιούμε το πλαίσιο EuroMed κατάρτιση, υποστήριξη επιθεωρήσεων, συντήρηση, συνολικός έλεγχος. Όπως είδατε βέβαια στα επίπεδα ασφαλείας, η ένταση της προσπάθειας εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Σε πράσινο έχουμε χώρες της Κεντρικής Αφρικής υπό το πλαίσιο FED, έργο που μας παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ζάμπια είναι ειδική περίπτωση. Είχαμε μια έκκληση προς στήριξη μέσω της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας. Έχουμε τις υποσαχάριες χώρες και τις δυτικές χώρες. Αυτά είναι προγράμματα που ε, αναμένουμε να εγκριθούν. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία εγκρίσεώς τους. γιατί οι ομάδες ελέγχων δεν, δεν ε, περνούν μόνο από τον ΕΑΣΑ, αλλά ε, χρειάζεται προσωπικό και από τις ίδιες τις χώρες, προκειμένου να έχουμε πλήρης ομάδες ελέγχου και επαρκές δυναμικό. Τώρα, πρέπει να αναπτύξουμε ε, κάποια στρατηγική προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί στη λειτουργία μας αλλά και στη σχεση κοστος κόστους-οφέλους. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να πάμε περίπτωση προς περίπτωση γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί οι πόροι που διατίθενται δεν είναι σε αντίστοιχο επίπεδο. Και έτσι αποφασίσαμε να πάμε περιφέρεια προς περιφέρεια ο ΕΑΣΑ ε, θεωρείται από, τον, από την ΙΚΑΟ ε, περιφερειακός οργανισμός ασφαλείας. Έχουμε τώρα έξι περιφέρειες στην Αφρική, αν ακούσαμε καλά τον ομιλητή, όπου καλύπτουν διάφορες χώρες. Μάλλον έχουμε έξι περιφερειακές οργανώσεις ασφαλείας στην Αφρική. όλα αυτά υπό την έννοια της αποτελεσματικότητας του κόστους ωφέλους. Άρα κάθε συντονιστής περιφερειακής ασφάλειας μας διευκολύνει συντονίζοντας στην οργανωτική μας προσπάθεια και όταν το έργο ολοκληρώνεται, αυτά που έχουμε παράσχει εν είδη έργου κατάρτισης μεθοδολογίας να μπορούν να είναι βιώσιμα. και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μια μόχλευση με τις περιφέρειες αυτές ώστε αυτά που θα έχουμε κάνει να μπορούν να συνεχιστούν. Θα έχουμε και την υποστήριξη που θα παρασχεθεί υπό το έργο EU Africa Safety and Aviation, EU ASA δηλαδή, για να εντοπίσουμε περαιτέρω κενά. Τώρα, να μην υπεραπλουστεύσω, αλλά έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής για τα βασικά πρότυπα ασφαλεία μόνο. Θα πρέπει να έχουμε διεθνώς έναν κλάδο αερομετοφορών που να είναι ασφαλής. Μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και οι αφρικανικές χώρες, βεβαίως, με την αυξημένη κυκλοφορία που υπάρχει στους εθέρες θα πρέπει να καταβάλουν όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια ελέγχου να αναλάβουν προσωπικό μεταξύ άλλων. Επίσης <clears throat> υπάρχει η απειλή των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Παρέχουμε λοιπόν υποστήριξη για αυτές τις νέου τύπου απειλές για την ασφάλεια Άλλο ένα ζήτημα πλέον είναι τα drones που βλέπουμε να κυκλοφορούν στους εθέρες όλο και πιο συχνά. Και στην Αφρική δεν βρίσκονται τόσα χρόνια πιο πίσω. Θα έχουμε όλο και περισσότερα τέτοια οχήματα αεροσκάφη στον αέρα. και θα πρέπει και αυτά να τα διαχειριστεί κανείς ε, σωστά. Και βεβαίω η πρόθεση της νέας τεχνολογία, <clears throat> κάτι που δεν είναι εύκολο για τις αφρικανικές χώρες και είναι μέρος των προτεραιοτήτων μας ή πρέπει να είναι. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξουν ε, επαρκείς επενδύσεις από τις χώρες αυτές προς την δορυφορική τεχνολογία και απλώς αναφέρω εδώ προγράμματα όπως τον Καλλιλέο, δηλαδή διορυφορικής πλοήγησης <clears throat> και στο πλαίσιο αυτό νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι και για το μέλλον ε, στο αφρικανικό πλαίσιο. Νομίζω ότι έχω φτάσει στο τέλος της ε, παρουσιασής μου και προτού ξαναδώσω στον Πίτερ το λόγο να αναφερθώ στη διαλειτουργικότητα, στη διασυνδεσιμότητα μάλλον, που είναι σημαντικός πολιτικός στόχος για τις αφρικανικές χώρες που μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν τα θεμέλια είναι υγιή. Εδώ το μήνυμα λοιπόν είναι να επαναλάβουμε και πάλι και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εσάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είμαστε ένα όχημα που επιτρέπει τη βελτίωση της ασφάλειας αλλά και την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στον αέρα. Ε, κάτι θέλετε να προσθέσετε, θέλετε, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλώς να συνοψίσω σε δύο-τρία σημεία την παρουσίαση που ακούσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ΆΖΑ και με την δική σας υποστήριξη προσπαθεί όχι μόνο να δει αν κινείται η σωστή κατεύθυνση η αεροπορική ασφάλεια στην Αφρική, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει κιόλα τον κλάδο όπου αυτό είναι δυνατό, ιδίω στα ζητήματα ασφάλεια. Θεωρούμε ότι η συνεργασία με την Αφρική είναι υποφελή και για τι δύο πλευρέ δεν ωφελεί μόνο τι Αφρικανικέ Αρχέ, αλλά και εμά του ίδιου εδώ στην Ευρώπη σε σχέση με όλη αυτή την αεροπορική ανάπτυξη που βλέπουμε στην Αφρικανική Ήπειρο. Και α μην ξεχνάμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε δυνατότητε συνεργασία και σε άλλου τομεί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες είναι ευγνώμονες για τη βοήθεια που τους δίνουμε στην ανάπτυξη της ασφάλειας ε, του αεροπορικού του κλάδου και όπως σας είπα ήμουνα σε μία συνεδρίαση του ΙΚΑΟ στην Ιγυρία και αυτό που έχω να πω είναι ότι ε, αν δεν αναλάβουμε εμεί το ρόλο αυτό θα τον αναλάβουν το ρόλο αυτό στον... στη δική μας τη θέση άλλη. Δίπλα μου καθόταν ένα εκπρόσωπο τη κινεζική αντιπροσωπεία και φάνηκε ότι ήταν έτοιμο να καλύψει οποιοδήποτε κενό θα άφηνε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση δηλαδή με τη συνεργασία στην Αφρική στον αεροπορικό τομέα. Μολονότι μπορεί να μην ακούγεται πολύ πολιτικά ορθό, μπορώ να πω ότι οι Αφρικανοί, οι Αφρικανοί προτιμούν να δουλεύουν μαζί μα, με του εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο πάντων, μπορεί να μην είναι πολύ πολιτικά ορθό, αλλά να το λέτε, αλλά είναι πολιτικά ορθό να το σκέφτεστε. Μαριάννα, δεν ξέρω αν ναι, εσύ έχει ε, κάποια σχόλια ή κάποιε ερωτήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, οι δύο αυτέ παρουσιάσει ήταν ιδιαίτερα πλήρη πολύ καλές. Μπορούμε να καταλάβουμε πλέον ποια είναι η δράση που έχει την αλάβει στην Αφρικανική Ήπειρο. Είναι σημαντικό να είναι ασφαλείς οι πτήσεις από την Αφρική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφρικανικές εταιρείες και να ρυθμίζονται και σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους επιβάτες αλλά τι γίνεται αντίστροφα όταν πετάμε από την Ευρώπη προς την Αφρική. Και αναφέρομαι στην ε, διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας, στη διαχείριση των αεροδρομίων. Ως προς αυτό τι κάνετε, πώς ε, χειρίζετε το ζήτημα αυτό, τι ελέγχους κάνετε, προκειμένου να παράσχετε την απαραίτητη ασφάλεια προς ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες εκτελούν πτήσεις προς την Αφρική. Από όσο ξέρω επίσης, δεν ε, υπάρχει σύστημα ιχνηλασιμότητας εντοπισμού των πτήσεων σε κάποιες ε, περιοχές της Αφρικής. Υπάρχουν ε, περιοχές της Αφρικανικής επικράτειας στις οποίες δεν καταφέρνουμε να εντοπίσουμε τις πτήσεις. Τι κάνουν προς αυτό. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, η ΆΖΑ, ουσιαστικά καταφέρνει να επιβάλλει στην Αφρική κάποια βασική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απουσία αφρικανικής νομοθεσίας. Βλέπουμε ότι αυτό ήδη συμβαίνει, το οποίο είναι πολύ θετικό. Τώρα, αναφερόμενοι στην Αφρική, πότε θα δοθούν ε, τα παρέτα χρήματα, ένα-δύο εκατομμύρια, προκειμένου να έχουμε την βάση αυτή που θέλουμε να κατασκευάσουμε στην Αφρική για το σύστημα έγνος. Μπορεί να μην συνδέεται άμεσα αυτό με τις αερομεταφορές, αλλά συνδέεται με το ζήτημα της αεροπορικής ασφάλειας. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. je Réponse... Euh, λοιπόν, ποιος θα απαντήσει σε ερωτήσει αυτές. Όσον αφορά τι υποδομέ αυτές που θέλουμε να έχουμε και στι δύο πλευρές για τις πτήσεις από και προς την Αφρική, βλέπετε ότι ο κύριος Μαρινέσου ασχολείται ιδιαίτερα με τα ζητήματα των αεροπορικών μεταφορών. Και βλέπουμε ότι ε, η Άζα χαίρει πολύ καλή φήμη στην Αφρική. αφού είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις σας, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις του κ. Μαρινέσκου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις αυτές όσον αφορά το πρώτο ζήτημα το οποίο θίξατε. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς προορισμού στην Αφρική και γίνονται και για αυτές προφανώς αξιολογήσεις ασφαλείας που ε, έμεσα μας δίνουν κάποιες πληροφορίες για τα προβλήματα που ενδεχομένω να αντιμετωπίζουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάλι θα αναφερθώ στην Ιγυρία γιατί είχα πάει εκεί πέρα πρόσφατα όπως σας είπα. Ο βασικός αεροδιάδρομος του Διεθνούς Αεροδρομίου στην Αμπούτζα άρχισε να εμφανίζει κάποιες τρύπες βασικά. Και ήταν οι αεροπορικές εταιρείες αυτές που είπαν στις αρμόδιες αρχές ότι δεν θα συνεχίσουμε να εκτελούμε πτήσεις αν δεν κάνετε τις απαραίτητες επισκευές στον αεροδιάδρομο. και τότε ανέλαβε μόνο δράση η κυβέρνηση, έκλεισε τον αεροδιάδρομο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακούστηκαν ε, πολλές αντιδράσεις βέβαια από το κοινό, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να επισκευάσει τον αεροδιάδρομο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι πληροφορίες που έχουμε από τις ίδιες αεροπορικές εταιρείε, από τους ίδιους τους αερομεταφορείς, μας βοηθούν να βελτιώσουμε το σύστημα ασφάλειας. Για το έγνος, ε, Έχετε απόλυτο δίκιο, πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα 5 εκατομμύρια όμως πρέπει να είναι το ποσό με το οποίο χρηματοδοτείτε. ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει και τις αφρικανικές χώρες να υποφεληθούν από αυτό, να χρησιμοποιείται περισσότερο το έγνος από τις αφρικανικές χώρες, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, πολλές φορές είναι το μόνο διαθέσιμο σύστημα το οποίο έχουν για να επιτηρούν και να εντοπίσουν να πάσα στιγμή και τις δικές τους αλλά και τις δικές μας, τις ευρωπαϊκές πτήσεις που πηγαίνουν προς την Αφρική. Προσπαθούμε λοιπόν με τα περιορισμένα μέσα που έχουμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα Ξέρετε ότι το πιο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε κάθε φορά να υποφελείται περισσότερο από όλη αυτή τη συνεργασία ο σύμβουλος εκείνος ο οποίος παράσχει την τεχνική υποστήριξη. Γι' αυτό το λόγο και εμείς ως ΕΑΖΑ θέλουμε να έχουμε τον γενικότερο σφαιρικό ρόλο επιθεώρησης της, εφαρμογή εφαρμογής του προγράμματος και το παρακολουθούμε έτσι καλύτερα και διασφαλίζουμε ότι όντως οι αφρικανικές χώρες γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Γιατί δεν θέλουμε απλώς να έχουμε επιτόπου στην Αφρική κάποιους συμβούλους μεσάζοντους ουσιαστικά οι οποίοι εποφελούνται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και λαμβάνουν αυτή τα εύσημα τελικά από τις αφρικανικές χώρες. Θα καταφέρουμε λοιπόν στο μέλλον και μελλοντικά προγράμματα να ενισχύσουμε περισσότερο το ρόλο αλλά και την προβολή της ΕΑΖΑ στην Αφρική για όλους αυτούς τους λόγους που σας εξήγησα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πρακτικής πλευράς, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο επιτόπου, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η φορεί παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα ανταποκρίνονται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέλουμε να υπάρχουν στην Αφρική. Αλλά βέβαια για αυτό το λόγο χρειαζόμαστε πολλούς πόρους. Δυστυχώς δεν τους έχουμε στην Άζα. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να προσλαμβάνουμε εμπειρογνώμονες από την ECI, από την ΑΙΑΤΑ, από την ΕΚΑΚ επίσης, προκειμένου να μπορούμε να παρεμβαίνουμε επιτόπου στις αφρικανικές χώρες, να μπορούμε να είμαστε δηλαδή επιτόπου και να επιβλέπουμε τελικά αν όντως οι απαραίτητες προδιαγραφές, τα απαραίτητα πρότυπα εφαρμόζονται. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι και οι ρυθμιστικές αρχές να καταλάβουν ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες του αεροπορικού κλάδου. Και πρέπει να συνδυάσουμε εδώ πέρα μια σειρά από μέτρα. Για να πάω όμως λίγο πιο πέρα στην ερώτησή σας, η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, Αφρικανική Νεπτυξιακή μάλλον Τράπεζα, κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα αυτό και αποφάσισαν ότι ε, θα πρέπει να παρέχουν και αυτοί τεχνικούς συμβούλους κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα για το οποίο απαιτείται μια χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα γίνεται στην περίπτωση αυτή του ε, αεροδιοδρόμου που παρουσίασε προβλήματα. Στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, πέρα από τη δική μας χρηματοδότηση, υπάρχει πλέον και η χρηματοδότηση από την Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Παράλληλα βέβαια έχουμε σαφώς και τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γενικά είναι πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι ε, επεμβαίνουν και όλοι μας προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ε, η ε, απαραίτητη ευκταία υποδομή όντως υφίσταται στην Αφρική και ότι όντως πληρεί τα πρότυπα ασφάλεια. Και για το έκνος να πω κάτι προς ενημέρωσή σας. Η ΑΣΕΚΝΑ που είναι μια ένωση 12 κρατών στην Αφρική αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το έγνος και όπως είπε και ο συναδελφός μου ο Πίτερ προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποια κίνητρα σε αφρικανικές αρχές για να επενδύσουν για αυτές περισσότερο στο έγνος και να χρησιμοποιούν τελικά το έγνος. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κριστίν έχει να κάνει ερωτήσεις, δεν θέλει το λόγο. Ο Μάριαν φαντάζομαι ότι έχει καλυφθεί από τις απαντήσεις που του δόθηκαν. Δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σε εδώ σήμερα. Μας διαφωτίσατε για ζητήματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια τη εβδομάδα αυτή που είναι αφιερωμένη στην Αφρική. Ξέρετε ότι πολύ συχνά αναφερόμαστε στον διεθνή ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροπορία. Μα δόθηκαν κάποια έμπρακτα παραδείγματα σήμερα τη διεθνού σα δράσης. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρουσία σα εδώ. στι 4 ε, Δεκεμβρίου 2017, στι 3 το μεσημέρι, είναι η επόμενη συνεδρίασή μα. Λύεται η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς.